Uh, uh, uh, Να ξεκινήσουμε αυτή την ακρόαση, σεμινάριο, συνεδρίαση, όπως θέλετε πείτε την. Να καλωσορίσω όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως τους προσκεκλημένους μας, τους εμπειρογνώμονές μας, που θα μας δώσουν πολλά στοιχεία και σημαντικές πληροφορίες. Στις 26 Απριλίου και εντός του γενικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε μια πρόταση για μια νέα οδηγία για την ισορροπία εργασιακής και οικονομικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται μετά την απόσυρση του 2015 της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις, για τις γονικές άδειες. Χαίρομαι πολύ που έχουμε οργανώσει αυτή την ακρόαση σήμερα, γιατί έτσι θα ξεκινήσουμε και τη δουλειά μας για αυτή την πρόταση της Επιτροπής εδώ στο ε, Κοινοβούλιο και στις ε, Επιτροπές μας και βεβαίως ε, προσβλέπω στις παρουσιάσεις που θα δώσουν σημαντικές πληροφορίες για την περαιτέρω εργασία μας. Να καλέσω τώρα τη συνάδελφο και συμπρόεδρο την κυρία Βίλγια Μπλικεβιτσιούτε που είναι από την Επιτροπή των ε, Γυναικών και της Ισότητας των Φίλων να μας ε, κάνει μια μικρή παρουσίαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο, την Μαρίτα Ουλσκοκ, για την εισαγωγή και για την οργάνωση της ακρόασης αυτής και την, ε, και την έμφαση που δίνει στην ισορροπία μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής μετά από αυτή την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως ε, πρέπει να ε, υποστηρίξουμε την ισότητα των φύλων, ε, υποστηρίζοντας την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες και οι άντρε πρέπει να γίνουν ίσοι και σε ό,τι αφορά τα εισόδηματα και σε ό,τι αφορά τη φροντίδα που παρέχουν. Και η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας έχει καταστεί ο πυρήνας της πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σήμερα η μεικτή αυτή ακρόαση θα επικεντρωθεί στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για τους φροντιστές και τους επίσημους και τους ανεπίσημους. 80% των ε, ε, αυτών σήμερα είναι γυναίκες. Ε, και βεβαίω η κατάσταση είναι ιδιαίτερως δύσκολη και του άτυπου φροντιστέ, γιατί η δουλειά του ούτε ρυθμίζεται ούτε καταγράφεται στα στατιστικά των κρατών μελών και συνήθω είναι μέλη οικογενείας άνθρωποι, και οι άνθρωποι που έχασαν την ε, δουλειά του. Οι φροντιστέ λοιπόν αυτοί δεν μπορούν να τύχουν κοινωνική προστασία, ούτε μπορούν να εξασκήσουν το δικαίωμα τη ισορροπία στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή και επίση είναι πολύ δύσκολο τομέα αυτό στη ρυθμισή του γιατί περισσότεροι από του φροντιστέ αυτούς κάνουν τη δουλειά τους σε ε, ιδιωτικές, ε, ιδιωτικά σπίτια όπου δεν μπορούν να μπουν οι ε, ελεγκτές εργασίας. Οπότε υπάρχουν δύο σχετικές εκθέσεις το 2016, μία για τις οικιακές βοηθούς, τις γυναίκες και μία για την ισορροπία επαγγελματικής οικογενειακής ζωής. Και οι δύο αυτές εκθέσεις μελετούν διάφορες πτυχές αυτού του εντελώς αρρύθμιστου τομέα εργασίας ο οποίος βεβαίως παίρνει όλο και περισσότερη σημασία στις ε, κοινωνίες μας, ακριβώς λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και των κοινωνιών μας. Επίσης, ε, για την, ε, στην έκθεση αυτή θα πρέπει να ζητείτε να υπάρξει προσαρμογή σε ευρωπαϊκά δεδομένα, έτσι ώστε κάθε γυναίκα ή άντρα να μπορεί να φροντίζει κάποιο, κάποιο μέλο τη οικογένειά του, χωρί όμω να πρέπει οπωσδήποτε να χάσει την δουλειά του. Επίσης να ε, του εγγυάμαστε κάποιο εισόδημα και κοινωνική προστασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει μια πρόταση οδηγίας για την, για την ισορροπία αυτών των δύο ειδών ζωής που δίνει τη δυνατότητα στις ε, γυναίκες να πάρουν πέντε μέρες το χρόνο άδεια ε, με πληρωμένη άδεια λόγω ασθενείας και χωρίς να χάσουν την ε, δουλειά τους. Δεν είναι πολύ, αλλά είναι μια καλή αρχή. Μια καλή αρχή μέσω αυτής της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση αυτή για τις οικιακές βοηθούς και τους φροντιστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση μελετά την ε, επισφάλεια των, ε, του καθεστώτος αυτού, του, αυτών των εργαζομένων, των φροντιστών, οι οποίοι πρέπει να ε, ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές κοινωνική ασφάλιση, υγείας και στην νομοθεσία για την αντιμετώπιση της ε, ε, της διακριτικής μεταχείρισης. Πρέπει να αναγνωριστεί ως πραγματική εργασία και αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης ε, της ε, παράνομης εργασίας θα μπορέσει να τους δώσει καλύτερη ισορροπία στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή τους. Εγώ έχω συνεργαστεί και για τις δύο αυτές ε, ε, εκθέσεις, οπότε πραγματικά καταλαβαίνετε πόσο με ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες που έχουμε προσκαλέσει. Πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Στέση Ιγκεμόνος, εκτελεστικό διευθυντή του Eurocarers. Έχετε 10 λεπτά για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Είναι τιμή μου να, είναι, να είμαι εδώ σήμερα. Αυτό που θα κάνω είναι να σας δώσω μια γενική κατάσταση των φροντιστών στην Ευρώπη, ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και ποια είναι η δική μας άποψη για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κοινωνικό πυλώνα. Καταρχάς για το δίκτυό μας. Το Eurocarers είναι ένα δίκτυο που συνδυάζει 70 μέλη και οργανισμούς τέρους από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Έχουμε 27 χώρες που εκπροσωπούνται στο δίκτυο. Οι μισές παρέχουν άμεσες υπηρεσίες στους φροντιστές, κατάρτιση, συμβουλευτική ενημέρωση και Επίσης ε, έχουμε και πολλές ε, ευρυντικέ δραστηριότητες ε, από ιδρύματα και πανεπιστήμια ώστε να έχουμε τα σχετικά δεδομένα. Επίσης έχουμε την γραμματεία ενός, μιας ομάδας συμφέροντος των Eurocares εδώ στο Κοινοβούλιο, οπότε σας ενδιαφέρει η κατάσταση των φροντιστών στην Ευρώπη και πώς μπορείτε να τους στηρίξετε, μπορείτε να γίνετε μέλη, έχω τις πληροφορίες αν θέλετε. Μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα είναι οι δημογραφικές αλλαγές που οδηγούν σε αύξηση των ε, ασθενειών που έχουν σχέση με την ε, ηλικία και Βεβαίω αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα συστήματα φροντίδα. Και αυτό ε, πιέζει πάρα πολύ και τι οικογένειε και τους άτυπους ε, φροντιστέ. Οι άτυποι φροντιστέ, ε, ο ορισμό τουλάχιστον που χρησιμοποιούμε εμεί, είναι αυτοί που παρέχουν αμυστή φροντίδα σε κάποιον που έχει μια χρόνια ασθένεια, μια αναπηρία ή οποιαδήποτε άλλη ανάγκη μακροχρόνια φροντίδα, εκτό επαγγελματικών πλαισίων. Οπότε μιλούμε κυρίω για γείτονε, για φίλου, για μέλη τη ίδια οικογένεια με το άτομο που χρειάζεται φροντίδα. Αυτό ξέρουμε για τους φροντιστές σήμερα με βάση τις ευρωπαϊκές έρευνες είναι ότι 80% της φροντίδας στην Ευρώπη παράσχεται από άτυπους φροντιστές. Και σύμφωνα και με τον ορισμό που σας ανέφερα πιο πριν, που είναι αρκετά ευρύς, το αναγνωρίζω, μιλάμε για 100 εκατομμύρια φροντιστές στην Ευρώπη. 20% δηλαδή του πληθυσμού της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Ένας ε, τυπικός ε, ε, φροντιστής είναι συνήθως μια γυναίκα μεταξύ 45 και 75 ετών. Η οικονομική τώρα αξία της άτυπης αυτής φροντίδας στην Ευρώπη, πάλι με βάση τις έρευνες, υπολογίζεται περίπου στο 50 έως 90% του, του συνολικού κόστους της επίσημης μακροπρόθεσμας φροντίδας. Επίσης έχουμε και κάποια εθνικά δεδομένα, όχι όμως για όλα τα κρατημένη δυστυχώς, να λοιπόν το πρώτο μήνυμα για εσά χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα, περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση των φροντιστών και το κόστος της φροντίδας στα διάφορα κράτη-μέλη. Γιατί βλέπουμε ότι αν οι φροντιστέ σταματήσουν αύριο να παρέχουν φροντίδα, το σύστημα απλώ θα καταρρεύσει. Οπότε, αν θέλουμε να του αντικαταστήσουμε, εν μία νυχτή θα πρέπει να δημιουργήσουμε είτε ένα νέο εκβάθρον σύστημα παροχή φροντίδα, ή, αυτό που θέλουμε εμείς, είναι να τους υποστηρίξουμε και να τους ενισχύσουμε. Αυτά γενικώ για την κατάσταση. Πέραν της γύρανσης του πληθυσμού, έχουμε και άλλους ε, ε, παράγοντες που επηρεάζουν ε, την κατάσταση, μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των συγγενών των οικογενειών, όλο και περισσότερες γυναίκες που μπαίνουν στην αγορά εργασία, το οποίο βεβαίως είναι καλή, θετική τάση, χαμηλές γεννήσεις, και ε, μεγαλύτερη διάρκεια εργασιακή ζωή. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν όλο και περισσότερη πίεση στις οικογένειες και στους φροντιστές. Εδώ βλέπετε έναν ε, ε, πίνακα, ένα γράφημα, μπορεί να μην βλέπετε απολύτω τι λεπτομέρειε, βλέπετε το πληθυσμό, το μέγεθο του πληθυσμού στην κάθε χώρα που ζει 25 χιλιόμετρα τουλάχιστον μακριά από την οικογένειά του. Πρόσφατα συνάντησα έναν ε, Έλληνα επαγγελματία που δουλεύει στο Λονδίνο, σε ένα πανεπιστήμιο στο Λονδίνο και μου είπε ότι ε, κάθε ε, Σαββατοκύριακο πρέπει να πηγαίνει πίσω στην Αθήνα για να φροντίζει τη μητέρα του η οποία όλη την εβδομάδα βρίσκεται σε έναν οίκο ευγυρία, αλλά το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει κάποιο να τη φροντίσει και ο άνθρωπο αυτό πηγαίνει μπρο πίσω στην Αθήνα και εδώ υπάρχει ένα γράφημα το οποίο μάλλον θα μπορείτε να διαβάσετε, οπότε το προσπερνώ. Ε, πέραν των όσων σας είπα πιο πριν, υπάρχει και η έλλειψη κάποιων ε, ε, επαγγελμάτων υγείας. Υπάρχουν ελλείψεις, πούμε, σε παθολόγους, σε φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους, φυσιοθεραπευτές η οποία είναι ουσιαστικά η ενδιάμεση μεταξύ της οικογένειας και του, ε, τομέα της, ε, του επίσημου τομέα παροχής ε, φροντίδας. Και υπάρχει βεβαίω και η σχετική ανακοίνωση ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μα δίνει τα σχετικά στοιχεία και χρονολογείται από το 2012. Τώρα, για τον αντίκτυπο τη άτυπη φροντίδα, όταν δεν υπάρχει στήριξη, υπάρχει περιορισμένη στήριξη που συμβαίνει σε πολλέ χώρε και πάλι με βάση τα ερευνητικά στοιχεία, βλέπουμε ότι πολλοί ε, φροντιστές αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν προσπαθούν να ε, συνδυάσουν τη δουλειά τους και την παροχή φροντίδας. Μπορεί να σας εκπλήξει αυτό, αλλά η, πλειοψηφία των φροντιστών προσπαθούν να κάνουν να έχουν ε, πλήρους απασχόλησης, απασχόληση. Αυτό σημαίνει ότι έχουν δύο ε, δουλειές πλήρους απασχόλησης και αυτό σημαίνει ιδιαίτερα προβλήματα, υψηλό κόστος και για τις εταιρείες και για την κοινωνία όταν πρόκειται να πάρει κάποιος άδεια ασθενείας και, αυτά, λοιπόν, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το βάλουμε στη συζήτηση. Επίσης ξέρουμε ότι άτυπη παροχή βοήθειας φροντίδας σημαίνει υψηλότερο κόστος για τους φροντιστές. Πολλοί εξ αυτών ε, συμβάλλουν στο κόστος της παροχής της φροντίδας. Και αυτό σημαίνει υψηλότερο κόστος για τους ίδιους και συνήθως τους οδηγεί στην φτώχεια ένα τρίτο των φροντιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, έχουν χρέη, ας πούμε. Και βεβαίω αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσει κανεί μια κοινωνική ζωή όταν, όπως είπα και πιο πριν, έχεις μια δουλειά πλήρους απασχόλησης και μετά έχεις να παράσχει και, έχει και φροντίδας. Τώρα, για την υγεία η πλειοψηφία των ε, φροντιστών ε, έχουν, ε, έχουν κατάθλιψη, είναι απομονωμένοι, αντιμετωπίζουν προβλήματα πνευματικής υγείας και πραγματικά είναι λίγο φαύλος κύκλος γιατί μετά αυτοί γίνονται ασθενείς οπότε το πράγμα διαιωνίζεται. Έχουμε διάφορα γραφήματα που το τονίζουν αυτό αλλά θα τα προσπεράσω αν μου επιτρέπετε. Τι θέλουν τώρα οι φροντιστές. Έγινε μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καταγράφει ε, με σειρά σημασία τις ανάγκες των ε, φροντιστών. Η πρώτη είναι η οικονομική στήριξη. Όπως είπα, πολλοί από αυτού. Ε, παρέχουν την βοήθεια αυτή, τη φροντίδα, χωρίς να έχουν καμία στήριξη και μάλιστα ε, δαπανούν και χρόνο και χρήμα και ενέργεια για να παράσουν τη βοήθεια, την ε, φροντίδα αυτή. Οπότε έτσι οδηγούνται σε πολλά προβλήματα. 42% των φροντιστών βρίσκονται στα χαμηλότερα εισοδήματα, δηλαδή δύο φορές το μέγεθος αυτών που δεν παρέχουν βοήθεια στην Ευρώπη. Η οικονομική στήριξη λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ε, ευέλικτες ε, συνθήκες εργασίας δεύτερον. Η πλειοψηφία των φροντιστών δεν επέλεξαν να γίνουν φροντιστές. Αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι κάποιος στην οικογένεια ασθενή και μια νυχτή βρίσκεσαι να πρέπει να του παράσχεις φροντίδα και πρέπει να αναδιοργανώσεις τη ζωή σου αναλόγως. Οπότε ε, ευέλικτες συνθήκες εργασίας και δυνατότητα παροχής άδειας είναι και αυτή στον, ψηλά στον κατάλογο. Επίσης, credits για την σύνταξη. Αν δούμε τη, την κατάσταση για την άτυπη παροχή φροντίδα στην Ευρώπη και το κενό, το συνταξιδοτικό κενό που υπάρχει, είναι επίσης πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη και το χρόνο που δαπανά κανείς να παράσχει βοήθεια όταν υπολογίζει ε, όταν υπολογίζεται η σύνταξή του. Επίσης, δυνατότητα σε ε, πρόσβασης σε ε, βοήθεια έτσι ώστε να αποφευθούν προβλήματα πνευματικής υγείας έτσι ώστε να σταματήσει να υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος. Και επίσης η κατάρτιση ή τέλος πάντων μια απλή πρόσβαση σε κάποιες βασικές πληροφορίες για το τι σημαίνει να είναι κανείς φροντιστής, ποιε είναι οι ασθένειε με τι οποίε πρέπει να, είναι, να έρθει αντιμέτωπο καθημερινά, κάποια υποστηρικτικά μέτρα ίσω που μπορεί να υπάρχουν ήδη στι χώρε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για του φροντιστέ να έχουν πρόσβαση σε αυτέ τι πληροφορίε. Και ακόμη και σε χώρε όπου υπάρχει επίπεδο καλό υποστηρικτικό, αυτέ οι πληροφορίε ε, δεν, ε, δεν, ε, οι φροντιστέ δεν έχουν πρόσβαση σε αυτέ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πολλά από όσα είπα αναφέρονται και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισορροπία Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής. Εμείς λοιπόν υποστηρίζουμε ένθερμα αυτή την πρόταση, θεωρούμε ότι είναι εξαιρετική, φυσικά δεν είναι τέλεια, τίποτα δεν είναι τέλειο. Θα μπορούσαμε κάποιες λεπτομέρειες να τις χτενίσουμε λίγο περισσότερο, αλλά νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για την αναγνώριση των φροντιστών, για την καταγραφή των φροντιστών, γιατί αν θέλει να υποστηρίξει κανείς τους φροντιστές πρέπει καταρχάς να τους αναγνωρίσει. Και σε πολλέ περιπτώσει αυτό δεν υπάρχει. Στην Ανατολική Ευρώπη, στι χώρε τη Μεσογείου δεν υπάρχει καν αυτή η δυνατότητα να καταγραφούν οι φροντιστέ. Οι πέντε μέρες ε, πληρωμένης ε, άδειας και άδειας ασθενείας επίσης. Η δυνατότητα της, ε, της πρόσβασης σε ευέλικτες συνθήκες εργασίας και η ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις στην επίσημη παροχή φροντίδας είναι πολύ σημαντικά. Η επιλογή είναι πολύ σημαντική και αυτό είναι, το, αυτός είναι ο πυρήνα ε, του μηνύματό μας. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την επιλογή να γίνουν φροντιστέ αν θέλουν, αλλά αν δεν θέλουν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κάποιες εναλλακτικέ λύσεις. Αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι ε, ε καλά στην πρόταση Κομισιόν. Τώρα για, τις, ε, για το διακανονισμό σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας, εδώ έχουμε κάποια επιθετικά σχόλια. Το έγγραφο δεν ε, περιγράφει επαρκώ πώς θα γίνει αυτό, πώς θα υπάρξει κάποιο είδους εποπτεία κτλ. Και βεβαίως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί γνωρίζουμε, όπως βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια, ότι ήδη Υπάρχουν κάποιες μεγάλες εταιρείες που ήδη παρέχουν ε, καλές υπηρεσίες στους ε, φροντιστές, στους ε, εργαζόμενους που έχουν και ευθύνε φροντιστού, αλλά βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει από όλους, ας πούμε δεν μπορεί να γίνει πολύ εύκολα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οπότε Καλό θα ήταν να εγκριθεί ο πυλώνα και η πρόταση αυτή, έτσι ώστε να μπορούμε να, ε, να ελέγξουμε πώ αυτό θα εφαρμοστεί για την περίπτωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τους χαμηλού εισοδήματος υπαλλήλου με επισφαλείς θέση εργασίας. Ας πούμε, θα είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι ε, εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτός ο πίνακας σας δείχνει και λυπάμαι αν δεν μπορείτε να το διαβάσετε, αλλά τα πράσινα τμήματα στον πίνακα δείχνουν το είδος των υποστηρικτικών μέτρων που υπάρχουν σε ευρωπαϊκά κρατημέλη. Καταγράφονται λοιπόν όλα τα υποστηρικτικά μέτρα στον πίνακα, όπω σα είπα, ε, ευέλικτε συνθήκε εργασία, κατάρτιση, πρόσβαση σε πληροφορίε και εισόδημα των ε, φροντιστών. Αν βλέπετε λοιπόν το πράσινο είναι θετικό. Αλλά αυτή είναι μια βασική μελέτη, πάντα ο διάβολο κρύβεται στι λεπτομέρειε. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν στι λεπτομέρειε είναι ότι χώρε με καλό υποστηρικτικό πλαίσιο συνήθως έχουν πολύ ε, περιοριστικά ε, πλαίσια. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι πάρα πολύ αυστηρά σε ό,τι αφορά το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε τέτοια μέτρα. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί, πολλοί φροντιστές δεν έχουν ιδέα ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοια υποστεκτικά ε, συστήματα. Επίσης, αν κάποιος έχει πρόσβαση σε ένα εισόδημα φροντιστού, αυτό είναι πάρα πολύ περιορισμένο, κάτω από το όριο της φτώχειας συνήθως. Η πολιτική προσέγγιση εκεί είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν θέλουν οι φροντιστές να παραμείνουν φροντιστές. Θέλουν να μπορούν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας, να κάνουν το φροντιστή για προσωρινό διάστημα. Αλλά βεβαίως πρέπει να υπάρχουν πάντα κάποιες εναλλακτικές. Το ίδιο ισχύει και για την σχέση μεταξύ του φροντιστού και του λαμβάνοντος τη φροντίδα. Σε κάποιες χώρες, ας πούμε, έχετε ε, πρόσβαση σε κάποια υποστηρικτικά μέτρα, αλλά μόνο αν ε, κάποιο από τα παιδιά σου είναι αυτό που χρειάζεται τη βοήθεια. Αν είναι ε, οι γονείς σου, δεν έχεις πρόσβαση σε τέτοια μέτρα. Για τι ευέλικτε συνθήκε εργασία. Αυτό πάλι επαφίεται στην διακριτική ευχαίρεια των εργοδοτών αν θα έχεις δηλαδή πρόσβαση σε τέτοιες ε, υποστηρικτικές ε, δομές ή όχι. Αυτό λοιπόν πρέπει να τυποποιηθεί λίγο περισσότερο. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν ε, πρόσβαση σε ένα βασικό επίπεδο στήριξης. Και θέλω επίσης να τονίσω και κάποιες καλές πρακτικές που ήδη υπάρχουν σε κάποιες εταιρείε. Το είδος των υποστηρικτικών μέτρων που υπάρχουν είναι πρακτικά μέτρα κυρίως ευέλικτες, ευέλικτο ωράριο εργασίας, ας πούμε. Αυτοί οι υπαλλήλοι που έχουν και ευθύνες φροντιστού συζητούν με τον εργοδότη τους και μπορούν να προσαρμόσουν λίγο το ωράριό τους χωρίς να πρέπει να χάσουν τη δουλειά τους. Ε, κάποια έκτακτη ας πούμε άδεια που πρέπει να πάρει ο φροντιστής μπορεί να αποζημιωθεί. Αυτό βέβαια κυρίω ισχύει για τις μεγάλες εταιρείε, γιατί είναι πιο εύκολο για αυτές. Πρέπει να ολοκληρώσω έτσι. Ναι. Ε, στήριξη που σχετίζεται με τη φροντίδα, ε, πρόσβαση σε εργαλεία, το ίντερνετ, η τηλέφωνα για να ψάξει κανείς για τις πληροφορίες, ε, συμβουλευτικές υπηρεσίες. Κάποιες εταιρείε ε, οργανώνουν τέτοιου είδους θεραπείες για τους φροντιστές και Βεβαίω πρέπει να περάσουμε και στο πακέτο τη, όλα αυτά πρέπει να περάσουν στο πακέτο για την ισορροπία τη οικογένειακή και τη επαγγελματική ζωή, Οπότε το συμπέρασμά μου και το αίτημά μα είναι το πακέτο για την ισορροπία τη επαγγελματική και οικογενειακής ζωή είναι πολύ καλό. Βεβαίω είναι ένα κομμάτι μια γενικότερη εικόνα. Χρειαζόμαστε το έγγραφο αυτό πρέπει να εγκριθεί γιατί ουσιαστικά αν οι φροντιστέ δεν υποστηριχθούν για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράσχουν καλής ποιότητας ε, φροντίδα σε καλές συνθήκες και να μπορούν να επιστρέψουν και στην επαγγελματική του ζωή, τότε τελικά αυτό θα σημαίνει ανάγκη σε μεγαλύτερε επενδύσει στα συστήματα φροντίδα και ξέρουμε αυτό ότι αυτό δεν μπορούν να το κάνουν τα περισσότερα κρατημέλη λόγω οικονομικών περιορισμών. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και βεβαίω προσβλέπω στην περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ηγημόνος για την παρουσίαση αυτή. Θα δώσω τον κύριο Κρίς Ουότερμαν το λόγο, πρόεδρο της Γεωπακόπα, για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να το πω στα Ιρλανδικά το κείμενο. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα, πιστεύω πως όχι. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω και εσάς και την Επιτροπή ΦΑΜ και την Επιτροπή Απασχόλησης που με καλέσατε και να σας πω πως παίρνω το λόγο σήμερα γιατί εκπροσωπώ εδώ την GIOPA που είναι μία οργάνωση που εκπροσωπεί όσους ε, οργάζονται στην γεωργία και στην ανθοκομία ε, γνωρίζετε την κόπα, εμείς εκπροσωπούμε τους ε, εργοδότες και έχει ξεκινήσει από το 1963 ο διάλογος μεταξύ εργοδοτών και συνδικάτων ε, για τα κοινωνικά θέματα στην Ευρώπη. Είναι πολύ δύσκολο η οικογενειακή ζωή και η επαγγελματική ζωή να συνδυαστούν. Και είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε μιλήσει πολύ το οποίο έχουμε συζητήσει πολύ με τα συνδικάτα. Και θέλουμε να δούμε και την πτυχή της γεωργίας και της ανθοκομίας σχετικά με το θέμα αυτό. Να σας πω δε πως υπάρχει το θέμα των συζύγων ανδρών και γυναικών που συνεργάζονται στα αγροκτήματά τους και κάνουν γεωργικές και ανθοκομικές εργασίες, όπως επίσης και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του γεωργικού κλάδου. Καταρχήν πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε ποιος είναι ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη σύζυγος. Εμείς ε, μέσω της Επιτροπής για την Ισότητα ε, βρήκαμε αυτό τον ορισμό που είπαμε εργαζόμενοι σύζυγοι είναι οι σύζυγοι οι οποίοι καταβάλουν εργασία στα πλαίσια ε, της ελεύθερης επαγγελματικής σχέσης ε, και όπου ε, συνεισφέρει μεν εργασιακά αλλά δεν αμείβεται απαραίτητος και πολύ συχνά δεν έχει και δικαίωμα σε κοινωνική προστασία και επιδόματα. Δηλαδή, ουσιαστικά καλύπτουμε τα γεωρικά αγροκτήματα, ε, τις ανθοκομικές εγκαταστάσεις όπου κάποιος από τους συζύγους εργάζεται μέσα αλλά δεν αμείβεται. Και αυτός που είναι ο κάτοχος ε, της, ε, του αγροκτήματος για παράδειγμα δεν αμείβεται με, ή δεν μισθοδοτείται αλλά ως ελεύθερος επαγγελματίας περιμένει να εισπράξει κάποια τιμολόγια. Μιλάμε δηλαδή για οικογενειακές επιχειρήσεις και οι περισσότερες αυτού του είδους στην Ευρώπη είναι ξεκάθαρα οικογενειακές όπου οι δύο σύζυγοι εργάζονται μαζί στο αγρόκτημα και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πάνω από το 90% της ε, εργασίας στο χώρο της γεωργίας στην Ευρώπη καλύπτεται από οικογενειακή εργασία. Αν δούμε τώρα τι κάνουν οι γυναίκες που έχουν τα δικά τους ε, αγροκτήματα ή οι δικές τους γεωργικές και ανθοκομικές επιχειρήσεις, τα στοιχεία της Eurostat από το θα μας πει το εξή μόνο το 30% των γυναικών έχουν στην κατοχή τους το ίδιο το αγρόκτημα. Είναι 3 εκατομμύρια γυναίκες λοιπόν που έχουν δικό τους αγρόκτημα ή ανθοκομική εκμετάλλευση. Και από τα στατιστικά στοιχεία γνωρίζουμε ότι το 57% των γυναικών που δραστηριοποιείται στην ανθοκομία και στη γεωργία είναι ε, σύζυγοι που βοηθούν τους σύζυγους τους στις εργασίες αυτές. Έχουμε όλο και περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες στην ανθοκομία και στη γεωργία, όπως και σε άλλους κλάδους, όμως δυστυχώς είναι πολύ λίγες οι γυναίκες οι οποίες έχουν τη δική τους αυτόνομη οικονομική δραστηριότητα και ο λόγος είναι η ανάγκη συμφιλίωσης της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής σε υπαίθριες περιοχές όπου δεν υπάρχει ε, κάποιο φροντίδα για τα παιδιά που είναι δύσκολη η πρόσβαση στην παιδεία, που είναι δύσκολη η πρόσβαση στην κατάρτιση. Ε, γιατί ξέρετε πως στην Ήπεθρο δεν είναι πάντα ίδιες οι δυνατότητες που προσφέρονται, όπως επίσης και η δυσκολία ε, στο να βρεθεί η, ε, η πίστοση, το δάνειο που θα σου επιτρέψει να στήσει τη δική σου επιχείρηση και αν χρειάζεται να δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες, 24 ώρες στη Γεωργία, ποιος θα φροντίζει τα παιδιά τους το Σαββατοκύριακο. Σήμερα πήρα το λόγο γιατί εκτός των όσων είπα προηγουμένως θα ήθελα να προσθέσω και μία ακόμα διάσταση που δεν είναι το πώς θα τους προσφέρουμε άδεια πατρότητα ή μητρότητας όταν γεννιούνται τα παιδιά. Δεν είναι μόνο το να βρεις κάποιον να φροντίζει τα παιδιά σου, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε πως ο ή η σύζυγος που ε, βοηθάει ε, ε, θα έχει δικαίωμα και στην κοινωνική ασφάλιση. Εγώ είμαι Βέλγος και μέχρι πρόσφατα οι σύζυγοι οι οποίοι εργάζονται στην επιχείρηση του άλλου σύζυγου είναι ανύπαρκτοι. Δεν πληρώνουν κοινωνικές εισφορές και το σύστημα δεν τους γνωρίζει. Και αν δείτε κάτω-κάτω στη διαφάνεια θα δείτε πως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως η κοινωνική προστασία ε, θα προσφερθεί ε, και στους συζύγους που ενεργοποιούνται στα συζυγικά αγροκτήματα, στην αδοκομεία, στη γεωργία, στα μικροκαταστήματα, στο λιανεμπόριο, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μέσω των δομών της ΚΟΠΑ εμείς κάναμε μία έρευνα. Στείλαμε δηλαδή ένα ερωτηματολόγιο στα μέλη μας, κράτη, στα διάφορα κράτη, και κάναμε μια σειρά ερωτήσεων. Για παράδειγμα, θελήσαμε να δούμε πώς έχει η κατάσταση εκεί και να σας πω περίπου τι τους ρωτήσαμε. Για παράδειγμα, στη χώρα σας αναγνωρίζετε νομικά το καθεστώς του ή της συζύγου που βοηθάει. Δεύτερον, εάν έχουν κάποιο είδους καθεστώ που αναγνωρίζεται, είναι υποχρεωτική η κοινωνική εισφορά ε, μέσω του συστήματος και αν όχι υπάρχει δυνατότητα αυτασφάλισης για παράδειγμα ή υπάρχει κάποιο άλλο είδος εθελοντικό σχέδιο ή καθεστώς μέσω του οποίου μπορεί να παρασχεθεί κάποιο είδος κοινωνική ασφάλιση στη χώρα σας. Έχετε κάποια δομή που επιτρέπει σε αυτόν της, το σύζυγο ή σύζυγο να αναπτύξει αυτές τις δραστηριότητες περαιτέρω, να λάβει κάποιο είδους επιδόματα ή βοήθεια έτσι ώστε να βοηθηθεί, να στηριχθεί και σε άλλες δράσεις. Έχετε βέλτιστες πρακτικές, θεωρείτε πως το καθεστώς αυτό είναι ικανοποιητικό. Και εδώ βλέπουμε ε, τις σημαίες ε, από τις χώρες από τις οποίες λάβαμε απαντήσεις, 12, 12 από τις 24 περιμέναμε και περιμένουμε να μας απαντήσουν κι άλλοι και πιστεύω πως τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα είναι και πολύ ενδιαφέροντα για τη δική σας Επιτροπή. Άρα λοιπόν για το κατά πόσο οι σύζυγοι που βοηθούν να αναγνωρίζονται νομικά με ένα δικό τους καθεστώς, δηλαδή αν ονομάζονται ε, κάπως και να αναγνωρίζονται κάποτε, είδατε πως 10 ναι, 2 όχι από τα κράτη που απάντησαν. Και εδώ θέλω να πω πως είναι σημαντικό να έχουμε και ένα ξεκάθαρο ορισμό του τι σημαίνει σύζυγος που βοηθάει. Γιατί είδαμε τα όσα έχουμε από το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φίλων στην Ευρώπη, αλλά δεν νομίζω πως ο ορισμός τους φτάνει. Γιατί αυτό που βλέπουμε σε πολλές χώρες είναι πως οι γυναίκες που ζουν στην Ήπεθρο μπορεί να έχουν ε, ας πούμε μια σύμβαση εργασίας που να καλύπτει 15 ώρο και να θεωρούνται εργαζόμενοι σύμφωνα με αυτό. Αλλά παράλληλα ε, να βάζουν άλλες 30 ώρες στο αγρόκτημα και να έχουν κοινωνική ασφάλιση για τις 15 ώρες που έχουν το συμβόλο και για τις 30 ώρες τις επιπλέον που κάνουν γεωργικές δουλειές να μην καλύπτονται και να μην υπάρχει και αυτό το καθεστώς ε, ε, εργαζόμενους, ε, υποβοηθ, μάλλον ε, συζύγου που βοηθάει, γιατί στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζονται μόνο ω εργαζόμενο για το 15ωρο και όχι για τις περιττέρω εργασίες που κάνουν υποβοηθητικά. Ε, ε υπάρχουν περιπτώσεις που αυτοί οι σύζυγοι που βοηθάνε έχουν και μια δεύτερη θέση εργασίας κάπου και μέσω αυτής ασφαλίζονται. Η δεύτερη λοιπόν ερώτηση είναι κατά πόσο ε, συνεισφέρουν, πληρώνουν κοινωνική ασφάλιση όταν έχουν αυτό το καθεστώ. Από τις 12 ερωτήσεις σε 8 χώρε είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν κοινωνική ασφάλιση. Σε δύο έχουμε θελοντικό καθεστώς και σε μία απάντηση είπαν υποχρεωτικό αλλά δεν πληρώνουν. Και μία χώρα όπου δεν χρειάζεται να πληρώσεις καθόλου ε, κοινωνική ασφάλιση. Όταν λοιπόν χρειάζεται να πληρωθεί θα, να καταβληθεί θα πρέπει να δείτε πώς υπολογίζεται αυτή. Σε κάποιες χώρες η υποχρέωση αυτή ε, να πληρωθεί ας πούμε εύκα ε, εξαρτάται όχι ή μάλλον βαρύνει όχι το ή σύζυγο που βοηθάει αλλά τον ή τη σύζυγο κάτοχο που θεωρείται εργοδότης. Οπότε το σημαντικό είναι πώς θα πληρωθεί αυτό το επιπλέον ποσό. Δηλαδή θα είναι επιπλέον στις κοινωνικές εισφορές που πληρώνει ο σύζυγος ή η σύζυγος που θεωρείται κάτοχος ή είναι ε, καλύπτεται ε, λόγω συζυγικής σχέσης. Είναι πολύ περίπλοκο. Και πολλές φορές αν χρειαστεί να πληρωθούν ε, οι εισφορές, ε, το σημαντικό είναι κατά πόσο, σε ποια βάση υπολογίζεται και αν ε, χρειάζεται κάποιο επιπλέον, κάποια επιπλέον εισφορά έτσι ώστε το επίπεδο να είναι αρκετά υψηλό. Δείτε λοιπόν εδώ τι, τι δικαιώματα και ε, προνοιακά επιδόματα καλύπτονται από αυτή την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Θα δείτε ότι σε κάποιες χώρες έχουμε κοινωνική ασφάλιση με δικαιώματα τα οποία είναι αυτά που βλέπετε στον κατάλογο. Αλλά πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί γιατί σε κάποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μπορεί κανείς να λάβει ε, ε, επιδόματα τέκνων, για παράδειγμα. Αλλά για τον σύζυγο. Οπότε εκεί χρειάζεται επιπλέον κοινωνική ασφάλιση, ε, που όμως δεν οδηγεί σε υψηλότερο επιδόματό τέκνου. Και αυτό συμβαίνει και σε άλλε περιπτώσει. Δηλαδή τα επιδόματα, παρόλο που μπορεί να πληρώνει επιπλέον κοινωνική ασφάλιση, δεν αυξάνονται. Άρα το κομμάτι ε, τη ε, επιπλέον κοινωνική ασφάλιση που πληρώνει ο σύζυγο ή η σύζυγο που βοηθάει, ουσιαστικά είναι άχρηστα. Γιατί δεν αυξάνουν τα επιδόματα τα οποία του δίνουν. Τώρα, για την Ιρλανδία έχουν ένα σύστημα εθελοντικών πληρωμών κοινωνική ασφάλισης, έτσι ώστε να δημιουργηθούν επιπλέον κοινωνικά δικαιώματα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορούσαμε να εξάγουμε και σε άλλες χώρες. Και το τελευταίο είναι, και το έχω ως ε, συμπέρασμα εδώ, ρωτήσαμε τα κράτη αν αυτό το καθεστώς του, ή ε, συζύγου που βοηθάει είναι ικανοποιητικό. Δεν θα σας πω ποιες ήταν οι χώρες που είναι ικανοποιημένες, αλλά πέντε δεν μας απάντησαν. Ή δεν ήταν σίγουρες. Οπότε υπήρξε ένα δισταγμό στο να απαντήσουν καταφατικά. Αυτό τι σημαίνει, ότι χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά ακόμα. Και συμπερασματικά να σας πω πως τέσσερα σημεία νομίζω από αυτά ε, στα οποία εγώ θα σταθώ κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρουν τη δική σας επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, επιπλέον των θεμάτων που συζητήσαμε, που είναι άδεια πατρότητας, μητρότητας, ε, φροντίδα για τα παιδιά. Εκτός από αυτά θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να προσφέρουμε κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνική ασφάλιση σε όλες αυτές οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται στη γεωργία και στην ανθοκομεία ως σύζυγοι και, κάνουν πολύ, και συνεισφέρουν πάρα πολύ. Θα πρέπει να γίνουν πιο ορατές και θα πρέπει να καλύπτονται από το σύστημα κοινωνικών παροχών. Σε όλα τα επίπεδα. Δεύτερον, πρέπει να εξετάσουμε πώς η συνεισφορά αυτή θα μετρηθεί, θα υπολογιστεί και πώς θα καταβάλλεται αυτή η εισφορά στο σύστημα. Δηλαδή, να δούμε αν μπορεί ε, αυτή η εισφορά να χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, ε, έτσι ώστε κάποια στιγμή να συνταξιδοτηθούν. Το τρίτο σημείο είναι η κοινωνική προστασία του ή της εργαζόμενης συζύγου. Είναι ένα θέμα που συνδέεται πολύ στενά με τη συμφιλίωση της εργασιακής και προσωπικής και οικογενειακής ζωής. Γι' αυτό σας καλούμε είτε στην επιτροπή, στις επιτροπές σας, είτε κάπου αλλού να ερευνήσετε το τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο με τους συζύγους που βοηθούν έτσι ώστε να λάβουμε 28 απαντήσεις αυτή τη φορά και να παροτρύνετε τα κράτη-μέλη που δεν έχουν τέτοιου είδους καθεστώς να το δημιουργήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βότερμαν. Θα δώσω τώρα το λόγο στην καθηγήτρια κυρία Κοτόφσκα από το Ινστιτούτο το Ινστιτούτο Στατιστικών και Δημογραφικών Θεμάτων από την Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Βασοβίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε το λόγο. Εγώ είμαι σε πολύ ευχα... στην πολύ ευχάριστη θέση να σας πω πως πολύ πρόσφατα τελειώσαμε μετά από ένα τριετές project για, τα... για την κοινωνία και τις οικογένειες. Και... και στα πλαίσια αυτού του προγράμματος έγιναν πολλές συζητήσει. Ε, στην τελική μορφή της έκθεσης διατυπώσαμε για κάποιες συστάσεις οι οποίες ε, συμβαδίζουν με την ε, οδηγία και όσο προβλέπει. Η οδηγία για την γονική άδεια λόγου χάρη δεν μπορεί να αναβάλλεται ιστοδυνικές. Πρέπει τώρα λοιπόν να ε, περάσουμε και να συζητήσουμε αυτή την πρωτοβουλία του Συμβουλίου. Για το ρόλο των συντάξεων βρίσκω το έγγραφο πολύ καλά διαρθρωμένο ως προς τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται. Εξαιρετικά επιχειρήματα για το, τι, για το λόγους, τους λόγους που μας κάνουν να χρειαζόμαστε αυτή την πρωτοβουλία. Όμως, είναι σημαντική και η προοπτική των οικογενειών, των οικοκυριών ως προς τα θέματα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας κάποια από τα πορίσματά μας. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η γονική άδεια και η άδεια των φροντιστών είναι σημαντικότατα στοιχεία για τη συμφιλίωση της ε, ε, εργασίας και της φροντίδας. Επίσης για την ισότητα των φύλων, την αγορά εργασίας και για την κοινωνική ισότητα μεταξύ ε, οικογενειών και ατόμων. Και θα ήθελα να αναπτύξω κάποια επιπλέον επιχειρήματα. Στο τέλος της ομιλίας μου θα ήθελα να εξηγήσω γιατί εμείς οι ερευνητές θεωρήσαμε αυτή την πρωτοβουλία μεγάλη σημασία. Κάποια από τα επιχειρήματα που θα ήθελα να σας παρουσιάσω ήδη αναπτύχθηκαν από τους συναδέλφους μου. Θα ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα πλέον. Βρισκόμαστε σε καιρούς όπου η οικογένεια αλλάζει. Όχι μόνο ως προς τις δημογραφικές τάσεις και δείκτες. Λιγότερα παιδιά, αστάθεια στην οικογενειακή δομή, ε, διαζύγια που είναι όλο και περισσότερα, διαφορετικές θεσμικές αλλαγές, λόγου χάρη μεγαλύτερη ποικιλία στις, στους σχηματισμούς των οικογενειών, στα οικογενειακά σχήματα που διαμορφώνονται, αλλά και δυσκολίες για την, οικογεν... για την επιβίωση της οικογένειας και την προσφορά της φροντίδας που χρειάζεται. Σε καιρού επισφαλών θέσεων εργασία και ανασφάλεια, το πρόβλημα του εισοδήματο είναι κεντρική σημασία. Νομίζω ότι η γυναικεία δουλειά, η δουλειά των γυναικών, η απασχόληση από την προοπτική μια οικογένεια είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι της οικονομικής αστάθειας της οικογένειας και λόγω των δυναμικών τάσεων στην αγορά εργασίας. Δεν μπορεί κανείς να παραμείνει εκτός αγοράς εργασίας για πολύ καιρό και να επανέλθει επιτυχώς όποτε, του, όποτε το επιθυμήσει. Όμως, όταν μιλάμε για το μακροπρόθεσμο ε, στοιχείο, εννοούμε μακροπρόθεσμα εισοδήματα. Για περισσότερο καιρό. Για την ε, για το καλό βιωτικό επίπεδο σε μεγαλύτερε ηλικίε. Αυτά πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε. Πώ θα συμφιλειώσουμε την δουλειά με την οικογένεια. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι όταν κοιτάζουμε την διάρθρωση τη κοινωνία ω προς την τρίτη ηλικία και τον αριθμό των ηλικιωμένων, αλλά και το πόσο πιο ανεξάρτητοι είναι οι άνθρωποι λόγω των πρόοδων της ιατρικής. Βλέπουμε ότι η ε, ανάγκη για φροντιστές αυξάνεται, όμως οι δυνατότητες των οικογενειών να στηρίξουν τους δικούς τους, να προσφέρουν αυτή τη φροντίδα, ε, μειώνεται όχι μόνο γιατί οι οικογενειακές δομές είναι πλέον λιγότερο ε, είναι, έχουν λιγότερα μέλη, αλλά και γιατί είναι αυτή η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Και όμω χρειαζόμαστε τις γυναίκες στην αγορά εργασίας, διότι ακριβώ υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά. Όλα αυτά αλληλοσυσχετίζονται. είναι αλληλένδετα και γι' αυτό πρέπει να τα δούμε από την προοπτική της αγοράς εργασίας. Πρέπει οι άνδρες να αναλάβουν ευθύνες ε, φροντίδας, όχι μόνο σε επίπεδο οικογένειας, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό. Γιατί θεωρούμε ότι η οδηγία αυτή είναι πραγματικά σημαντική. Μια σημαντική πρωτοβουλία. Πρώτον, Έχουμε κάποια αποτελέσματα σε ένα επίπεδο μικροστατιστικής από έρευνες που εξήγαμε σε διαφορετικές χώρες με ποιοτικά και ποσοτικά ε, στοιχεία και είδαμε ξεκάθαρα τα αποτελέσματα αυτά ότι σε επίπεδο οικογενείας είναι πολύ σημαντικό η ιδιότητα του πατρός, ο ρόλος των ανδρών να ε, γίνεται αντιληπτός ως ένας κοινωνικός ρόλος, όχι απλώς ως ένα δικαίωμα ή ως ένα προνόμιο. Δηλαδή αλλάζει η αντίληψη για τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών στην οικογένεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση και προς τα εκεί πρέπει να στραφούμε. Και από τις ποιοτικέ μας μελέτες ε, εξήβραμε ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις στις οικογένειες ότι η άδεια πατρότητας θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή, όχι ως ευκαιρία προς εκμετάλλευση, αλλά ως ένα δικαίωμα κοινωνικό που οφείλεται να ασκείται. Τώρα για την αντίδραση των εργοδοτών, των εταιριών στο να αναλάβουν αυτή την ευθύνη της γονικής άδεια ε, που θα δείτε και, δίδεται και στους πατεράδες. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ξεκάθαρα ότι όταν υπάρχει εξατομικευμένο δικαίωμα στη γονική άδεια, μπορεί να θεωρηθεί καλύτερο μέτρο για να πιστούν και οι εργοδότες ότι πρέπει να το παραχωρήσουν. Είναι ευκολότερο δηλαδή να μπορέσουν οι πατεράδες να χρησιμοποιήσουν τα μέτρα του κανονισμού εφόσον περάσουν έτσι. Αλλά να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η γονική άδεια έχει και θετική επίπτωση στον οικογενειακό βίο. Πρώτα απ' όλα, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις σκανδιναβικές χώρες ε, περί γονικής άδειας, εκεί όπου η γονική άδεια έχει θεσπιστεί εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε αρκετά μακροχρόνια ε, δεδομένα για να δούμε πώς έχει διοργανωθεί η οικογενειακή ζωή, βλέπουμε ότι η άδεια πατρότητας, ιδίως για το πρώτο παιδί, σχετίζεται με την ε, θετική ε, έκβαση και την διάρκεια στον χρόνο της ένωσης. Λιγότερες εντάσεις στην οικογενειακή ζωή. Και έχουμε και ποσοτικά δεδομένα γι' αυτό. Ταυτόχρονα υπάρχουν αποδεκτικά στοιχεία ότι διευκολύνεται και η μετάβαση στο δεύτερο παιδί. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι και ένα μέτρο για να χρησιμοποιηθεί και να μπορέσουν οι γονείς να εκπληρώσουν τις γονεϊκές τους προσδοκίες, τις φιλοδοξίες τους, δηλαδή να έχουν οικογένεια με την υπογεννητικότητα να σώβει στην Ευρώπη. Όσον αφορά τη φροντίδα προς τους ηλικιωμένους, αυτά τα μικροστατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι η οικογένεια θεωρείται ακόμη ως σημαντικότατη πηγή φροντίδας. Ακόμα και οι εργαζόμενοι, αυτοί που είναι ειδικοί στην αγορά εργασία, συμμετέχουν στη φροντίδα. Και οι πιθανότητες να ασχοληθούν με τη φροντίδα για τους ηλικιωμένου είναι πολύ ψηλή, πολύ μεγάλη για, την, ε, για τους εργαζόμενους. Η πενθήμερη άδεια για σκοπούς φροντίδας είναι απλώς ένα πρώτο βήμα για να υπάρχουν ακόμη ευρύτερα μέτρα, διότι πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει και παράταση του επαγγελματικού βίου. Ε, μιλάμε για ανθρώπους μεταξύ των 45 και των 70-75. Πόσο να παραμένουν στην αγορά εργασίας. Οι συνέπειες είναι θετικές λοιπόν και σε επίπεδο οικογένειας, αλλά συμβάλλει και στο να υπάρχουν ακόμη περισσότεροι εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας. Και τελευταίο, τέλος, ε, ότι να πω ότι κοιτάξαμε τα εκτελεστικά μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν την επιλογή του ενός ή του άλλου μέτρου. Δηλαδή, υποβάλλοντας κάποια πρόταση, μπορεί να διαμορφώσουμε τις συμπεριφορές των ανθρώπων, τις προσδοκίες τους και τις συμπεριφορές τους. Η αλλαγή στην αντίληψη για το τι είναι συμμετοχή του πατέρα στην φροντίδα λόγου χάρη, ή αν θέλουμε να μιλάμε για ίση κατανομή των ευθυνών ως προς το εισόδημα έχουμε ήδη μια πολύ καλή λύση. Στο τέλος της παρουσίασής μου ήθελα απλώς να σταθώ σε αυτή τη δήλωση της τελικής μας έκθεσης που αναφέρει ότι ελπίζουμε και περιμένουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αναβάλουν άλλο την εξέταση αυτών των θεμάτων και να ε, εκπληρώσουν τις προσδοκίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα να σας απευθυνθώ. Ευχαριστούμε πολύ την καθηγήτρια Ιρένα Κοτόφσκα και τώρα λόγο στην κυρία Πάολα Παντζέρη, η οποία είναι υπεύθυνη για θέματα ε, συμβουλευτικής προσκογένειας ε, και ε, σας δίνω 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα να σας απευθυνθώ σήμερα και να σας παρουσιάσω την άποψη της Κοφάσε οικογένειες της Ευρώπης για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Θα ήθελα σήμερα να σας εξηγήσω ποιοι είμαστε σε περίπτωση που δεν μας γνωρίζετε και να παρουσιάσω τις θέσεις μας για την εξισορρόπηση επαγγελματικού και οικονομικού βίου και ιδίως για τους φροντιστές. Η ΚΟΦΑΣΕ, η Οικογένεια τη Ευρώπη, είναι μια πολυφωνική οργάνωση με 60 οργανωσμούς να συμμετέχουν από 24 κάτι μελη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδρυθήκαμε το 1958 ένα χρόνο μετά τη συνθήκη της Ρώμης. Μεγαλώνουμε ταυτόχρονα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτούμαστε κυρίως από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Κοινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύνθημά μας, το μότο μας είναι μια καλύτερη κοινωνία για όλες τις οικογένειες. Και βεβαίω η εξισορρόπηση επαγγελματικού και γενικού βιού είναι από τι βασικέ προτεραιότητε όλα τα μέλη μα για να πετύχουμε καλύτερη ζωή για όλε τι οικογένειε. Εργαζόμαστε σε μια σειρά από διαφορετικούς τομείς, θεματικούς τομείς. Ελπίζω να τα βλέπετε από την παιδεία μέχρι την ισορροπία ζωής ιδιωτικής και επαγγελματική μέχρι τα δικαιώματα καταναλωτών. Προσπαθούμε να κάνουμε τη φωνή των οικογενειών να ακουστεί μέσα στην ποικιλομορφία του σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να δούμε τι ακριβώς κάνει η Ευρώπη για τα μέλη μας. Ό,τι αφορά την ισορροπία ε, επαγγελματικού και οικογενειακού βίου να υπογραμμίσω την προσέγγιση που έχουμε ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια. Σα έχω βάλει εδώ μερικά κομμάτια πάζλ, γιατί κάθε οικογένεια είναι διαφορετική και κάθε οικογένεια έχει διαφορετικέ ανάγκε. Δεν υπάρχει μια κοινή λύση για όλου για να συμφιλειωθούν επαγγελματικώ με τον οικογενειακό βίο. Πρέπει κάθε οικογένεια να έχει ένα δίχτυ ασφαλεία μέτρων. Μια σειρά μέτρων που μπορούν να αναλυφθούν ώστε να καλυφθούν συγκεκριμένε ανάγκε μια δεδομένη οικογένεια όταν μιλάμε για φροντίδα ενό παιδιού, ενό ηλικιωμένου γονέα, ανθρώπων με αναπηρίε που μπορεί να είναι μέλη τη οικογένεια. Και την προσέγγιση αυτή την ονομάζουμε αρεστή. Πόροι, υπηρεσίε, χρόνο. Η οικογένεια πρέπει να έχει αρκετού πόρου, δικαιότερα φορολογικά συστήματα λοιπόν, οι καλύτερα εισοδήματα για να μπορούν να έχουν μια εξωτερική ζωή, ή υπηρεσίε, υπηρεσίε φροντίδα ε, για τα παιδιά, για του ηλικιωμένου, για παιδιά με αναπηρίε, που χρειάζονται έκτακτη ιατρική φροντίδα και χρόνο. Χρόνο για να μπορούν να είναι μαζί. Χρόνο άδεια ή ευέλικτου διακανονισμού στην εργασία. Και αυτά καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωή. Η εξισορρόπηση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου πολύ συχνά βιου πολυ αντιληπτή ω ένα προνόμιο για τι νέε μητέρε που μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά του. Αυτή η προσέγγιση αλλάζει, αλλά και πάλι είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε ότι η ισορροπία επαγγελματικού και γενοβίου πρέπει να καλύπτει όλο το φάσμα τη ζωή. Δεν είναι ένα προνόμιο για τι νέε μητέρε. Δεν είναι επίδομα. Είναι κάτι που όπω σωστά αναφέρατε στο ψήφισμά σα του Σεπτεμβρίου, είναι ένα δικαίωμα για όλου η ισορροπία επαγγελματικού οικογενειακού βίου. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια διάσταση του φύλου, όπω αναφέρθηκε προηγουμένω ω προ τη φροντίδα, και υπάρχει και η γενιά σάντουιτ. Όλο και περισσότερο γυναίκε των 45-50 και άνω πρέπει να ασχολούνται με παιδιά, ε, χωρί να είναι αναγκαστικά ε, ε, ανεξάρτητε οικονομικά. Πρέπει να ασχολούνται λοιπόν με παιδιά, εγγόνια ή γονεί και πεθερικά. Όχι μόνο του δικού του γονεί και όλα τα πεθερικά του. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Ευρωπαϊκή ολα τα πεθερικα του οπω αναφερθηκε προηγουμενω η ευρωπαικη επιτροπη πρότεινε ένα πακέτο για την εξισορρόπηση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου στι 26 Απριλίου, που αποτελείται από μια οδηγία και μια ανακοίνωση. Ένα συνδυασμό νομοθετικών και μη νομοθετικών προτάσεων για να αρχίσει αυτή η αλλαγή. Επίση, αυτό έγινε κατόπιν αιτήματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ένα ψήφισμα του περασμένου Σεπτεμβρίου, το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά τον συνεισηγητή τον βασικό μελλον εισηγητή. Εδώ να πούμε ότι ένα από τα θέματα που ε, άγγιζε το ψήφισμα ήταν οι φροντιστέ και είναι πολύ, σωστός, πολύ σωστή κατεύθυνση που επελέγει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλαβε τα αιτήματά μα και πρότεινε μια συγκεκριμένη δράση, κίνηση για να επιληφθούν και άλλα προβλήματα των οικογενειών. Τώρα, η δική μα άποψη συνοψίζεται στο εγγραφό Families on the Edge. Οι, γυναίκες, οι, οι οικογένειε ε, τα πρόθυρα κρίσης. Ε, εδώ Δίνουμε όλες μας τις απόψεις για το τι συμβαίνει σήμερα στις οικογένειες και μια λεπτομερή αποτίμηση του πακέτου για την εξισορρόπηση οικογενειακού ε, επαγγελματικού βίου. Όπως είπε και η συνάδελφος, και εμείς πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή, το πακέτο αυτό είναι μια καλή πρόταση, διότι ακολουθεί μια σωστή νομική άποψη, δίνει δυνατότητα στην Ευρώπη να δείξει τον ανθρώπινο πρόσωπό τη και να, δει, να φέρει αλλαγέ στη ζωή των πολιτών, στου κατοίκου τη Ευρώπη, σε όσου διαμένουν εδώ. Είναι μια χειροπιαστή προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά ελπίζουμε η πρόταση αυτή να περάσει χωρί να μπλοκαριστεί ή να αποδυναμωθεί ή να μην κολλήσει σε ιδεολογικέ συζητήσει. Δεν είναι θέμα ιδεολογία αυτό. Είναι κάτι που το χρειάζονται οι οικογένειε και είναι κάτι που πρέπει να του δοθεί και γρήγορα. Στην αποτίμησή μα καλύπτουμε και την οδηγία και την ε, ανακοίνωση και θα προσπαθήσουμε μια-δυο διαφάνειε να σταθώ στη διάσταση των φροντιστών. Έχουμε τρει βασικέ πτυχέ που αφορούν του φροντιστέ. Πρώτα απ' όλα ε, οι υπηρεσίες, μετά οι δεξιότητε και τρίτον τη διακανονισμοί στην εργασία. Αυτά χρειάζονται οι φροντιστές. Πρώτα απ' όλα για τι υπηρεσίε. Το να στηρίξουμε του φροντιστέ είναι να του παρέχουμε και υπηρεσίε για την ενεργό ε, συμπερίληψη και την καλή διαβίωση των ανθρώπων που είναι φροντιστέ ή παρέχουν φροντίδα και όσων τη δέχονται. Δεν χρειάζεται δηλαδή απλώ να βγάζουμε ανθρώπου στην αγορά εργασία για να παρέχουν φροντίδα, αλλά να μένουν στην αγορά εργασία. Θέλουν οι άνθρωποι αυτοί να παραμένουν σε θέση εργασία και να παρέχουν φροντίδα. Φροντίδα σε επίπεδο κοινότητα ίσω. να βασίζεται στι ανάγκε τη κοινότητα. Ε, υπηρεσίε ποιότητα. υπηρεσίε δεν μπορεί να είναι ε, μη ποιοτικέ, γιατί καμία οικογένεια δεν θα δεχτεί ένα εξωτερικό που δεν παρέχει υπηρεσίε ποιότητα να τα παρέχει. Επίση, να είναι και η εγκύτητα ένα κριτήριο και η τιμή. Εάν η τιμή είναι πολύ ψηλή, η οικογένεια θα ε, σταματήσει να δουλεύει. Πώ μπορεί να σταματήσει να δουλεύει όμω όταν πρέπει να παρέχει ταυτόχρονα και φροντίδα και να καλύπτει την υψηλή τιμή. Εδώ μπορεί να διαδραματιστεί πολύ σημαντικό ρόλο από το Γενικό Ταμείο. Ε, πρέπει να, να προβλεφθεί η υποδομή, το δίκτυο και η διάρθρωση ε, για τους φροντιστές. Πολλά έχουν γίνει ως τώρα, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερο ώστε και στο επόμενο διάστημα προγραμματισμού να προβλεφθούν κονδύλια για την εξισορρόπηση επαγγελματικού και γενικού βίου. Επίσης υπάρχει κάτι που το ονομάζουμε στόχο για τη φροντίδα πέραν τη φροντίδα των παιδιών. Υπάρχουν σχετικοί στόχοι τη Βαρκελόνη στα πλαίσια αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να σκεφτούμε τώρα την εκπόνηση δικτών πέρα τη φροντίδα των παιδιών. Εδώ δείκτη αξιολογική ε, σύγκριση είναι σημαντική για όλε τι μορφέ φροντίδα, για όλε τι μορφέ υπηρεσία που παρέχονται. Δεν χρειάζονται όλοι τα ίδια, ούτε όλοι θα υποφεληθούν από την προσφορά μια υπηρεσία, εάν είναι ολόιδιε οι προσφορέ όλη την Ευρώπη. Είναι διαφορετικέ οι αυτό έχει να κάνει και με την κατοίκο ε, υποστήριξη. Υπάρχουν κάποια είδη φροντίδα ε, και υποστήριξη που μπορούν να παρασκευθούν στα πλαίσια μια κοινότητα κατοίκων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου στην προσέγγιση μα. Επίση, να τονίσω ότι οι υπηρεσίε στήριξη για του φροντιστέ δεν θα πρέπει να γίνονται αντιληπτέ ω ένα εργαλείο να μείνουν οι άνθρωποι στην αγορά εργασία. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι κάτι που θα του επιτρέπει, επιτρέπει στα μέλη οικογένεια να παραμείνουν σε ε, αμοιβόμενη εργασία αλλά είναι ένα σύστημα που θα χρησιμοποιήσει κυρίω του χρήστε, αυτού που πραγματικά χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε. Με κοινωνική, ενεργή συμμετοχή και ανεξάρτητη ζωή. Τελευταίο σημείο, μια διαδικασία ε, παρακολούθηση τη πρόοδου μέσω τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμένου. Ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμενο έχει τεράστιο αντίκτυπο στο πώ εκπονούνται οι πολιτικέ στα κράτη-μέλη. Χρησιμοποιείται για να παρακολουθούνται ε, και να καταμετράται η πρόοδο στα μακροχρόνια στον τομέα τη φροντίδα. Εδώ επικεντρώνομαι στου φροντιστέ επίπεδο οικογένεια, αλλά να τονίσω το εξή σε κάποιε χώρε η έλλειψη υπηρεσιών είναι τόσο μεγάλη που είναι πολλέ οι μετανάστευε, μιλάμε για εκατομμύρια γυναίκες, προσλαμβάνονται και απασχολούνται ως φροντιστές ε, σε πλήρη απασχόληση. Πολλέ φορές ζουν ε, σε, ε, σε άλλη χώρα, πολλέ φορές καλύπτουν απλώς το κενό του κράτους πρόνοια που δεν υπάρχει. Και Μπορεί να μην είναι στην οικογένεια, αλλά θα πρέπει να έχουν και εκείνε ε, ε, ισορροπία επαγγελματικού και γενιακού βίου και τι σωστέ αμοιβέ. Μην το ξεχνάμε, αυτό συμβαίνει καθημερινά σε πολλά σπίτια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αναγνωριστεί. Για να προχωρήσουμε, τα συστήματα αυτά για τη στήριξη των φροντιστών, επιτρέποντα να παραμείνουν σε αμοιβόμενη θέση εργασία, ενώ έχουν το χρόνο να παρέχουν και φροντίδα για τα μέλη τη οικογένεια του, είναι σημαντικό. Πρέπει να καλωσορίσουμε και την πρόταση τη σύντομη άδεια για φροντιστέ, την πενθήμερη αυτή άδεια που προτείνεται με αμοιβή, ε, να πούμε ότι θα ήταν καλύτερο να είναι παραπάνω από πέντε μέρε βέβαια, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να διαβρύνουμε τον ορισμό για την επιλεξιμότητα των φροντιστών. Δεν είναι μόνο οι συγγενεί πρώτου βαθμού σε ένα πλαίσιο τέτοια κινητικότητα όπου οι οικογένειε που ξεπερνούν τα σύνορα των χωρών, ε, η κινητικότητα των εργαζομένων επιβάλλει τέτοια κυκλοφορία, αλλά πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα αδέρφια και οποιονδήποτε άλλο επιλέξει αυτό που χρειάζεται φροντίδα ω φροντιστή. Υπάρχουν κατάλληλα άτομα που μπορεί να μην είναι Αναγκαστικά οι γονεί μπορεί να είναι φίλοι γείτονε, ανάλογα με τη μορφή τη φροντίδα που παρέχεται. Επίση, θα πρέπει να χαρτογραφηθούν οι ανάγκε για τι ε, ανάγκε αδειών για φροντιστέ μακροπρόθεσμα. Ε, υπάρχουν επικουρικέ φροντίδε, να τα σκεφτούμε και αυτά. Στο μέλλον, ίσω πρέπει να σκεφτούμε όχι αναγκαστικά σε αυτή την οδηγία, αλλά μελλοντικά. Να προβλέψουμε ένα σύστημα για να καλύψουμε και αυτέ τι ανάγκε. Τέλο, οι ευέλικτοι διακανονισμοί εργασία. Νομίζουμε ότι είναι πολύ θετικό μέτρο αυτό που συμπεριλήφθη στην πρόταση της οδηγίας και θέλουμε να υπάρχουν τέτοιοι ευέλικτοι διακανονισμοί και για τους φροντιστές. Όμω, να απευθύνουμε έκκληση για την αιτιολόγηση τη άρνηση γραπτό, για να είμαστε βέβαιοι ότι τα μέτρα αυτά τα παίρνουν σοβαρά οι εργοδότε. Επίση, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε ότι ένα αριθμό μορφών ευέλικτων διακανονισμών για την εργασία ήδη αναφέρονται και έχουν εισαχθεί όχι μόνο η μείωση των ορών, αλλά και η αλλαγή των μορφών εργασία και η χρήση τη ε, τηλεεργασία ή τη εφηού εργασία. Ένα κίνδυνο που θέλουμε να τονίσουμε εδώ είναι ο κίνδυνο να περάσουμε από την οτροπία τη παρουσία στη δουλειά, τη ε, νοοτροπία τη διαθεσιμότητα. Όταν μιλάμε για ευέλικτη εργασία και θέλουμε να δώσουμε αυτό το δικαίωμα, θα πρέπει να σκεφτούμε και το δικαίωμα τη αποσύνδεση. Δηλαδή, πού σταματάει η ευελιξία και πού αρχίζει ο οικογενειακό βίο. Πότε είναι κανεί διαθέσιμο και πότε δεν είναι. Να απαντάω σε ένα email μέσα στα μεσάνυχτα, ενώ έχω γυρίσει σπίτι μου, α πούμε. Θα το περάσω αυτό, αλλά για την εκστρατεία ενημερώσεις, που τώρα εξάγουμε, μια μελέτη για τις ανάγκες των φροντιστών ε, των οικογενειών. Ε, σε οκτώ γλώσσες είναι διαθέσιμο στο ίντερνετ. Ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, πορτογαλικά, σλοβενικά, ισπανικά. Είναι ανώνυμη η μελέτη. Μπορείτε να τη συμπληρώσετε online. Παίρνει λίγα μόνο λεπτά. Αυτό είναι το link, ο σύνδεσμος Μπορώ να σας δώσω και άλλα στοιχεία, αλλά δείτε τα και στο website, ε, είναι ακόμα ανοιχτή η μελέτη. Έχετε το δικαίωμα λοιπόν εδώ να εκφράσετε τη δική σας άποψη, εκμεταλλευτείτε την. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Τώρα μπορούμε να ακούσουμε τα μέλη, να ακούσουμε σχόλια, ερωτήσεις. Ο κύριος Σόκορ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέκερ μου ζήτησε να παρέμβω εκ μέρους του γιατί δεν μπορεί να είναι εδώ και θέλω κι εγώ να κάνω κάποια σχόλια. 70% ε, των ε, φροντιστών στην Ευρώπη είναι φίλοι ή μέλη της οικογένειας. Άνθρωποι που φροντίζουν τις οικογένειές του συνήθως είναι οι γυναίκες. Πολλοί αφήνουν τη δουλειά τους για να φροντίσουν το μέλλον της, το οικογένειας που έχει ανάγκη η φροντίδα. Αυτό έχει επιπτώσει και στην ε, αγορά εργασία και στο εισόδημά του, αλλά και στην φυσική και πνευματική του υγεία. Οι φροντιστέ αποτελούν ένα ραχοκοκαλιά του συστήματο φροντίδα στην Ευρώπη και γι' αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε τη δουλειά και τι θυσίε που κάνουν. Χρειάζεται ισχυρή φωνή για του φροντιστέ στην Ευρώπη. Περισσότερο ευέλικτε ώρε εργασία μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη ισορροπία επαγγελματικού και οικογενειακού βίου για τι οικογένειε στην Ευρώπη. Καλωσορίζουμε την πρόταση Κομισιόν για την ισορροπία αυτή και την ε, συμπερίληψη τη ε, πενθήμερη άδεια αναέτος, αλλά και της ε, δυνατότητας ε, ε, ευέλικτων ωραρίων εργασίας και προσαρμογής του ωραρίου εργασίας. Οι φροντιστές δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να αφήσουν την δουλειά τους, αλλά θα πρέπει καλύτερα να μπορούν να ισορροπήσουν την εργασιακή και την οικογενειακή του ζωή. Είναι σημαντική λοιπόν η συμβολή των ανθρώπων αυτών στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Και επίσης να προσθέσω εγώ στα όσα λέει ο κύριος Μπέκερ για τις ε, αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η οδηγία των, ε, των αποσπασμένων εργαζομένων ε, σε όσους όντως χρειάζονται βοήθεια. Από όσο ξέρω, στη Γερμανία πάνω από 200.000 οικογένειες εξαρτώνται από την ε, ε, παροχή φροντίδας από τα ίδια τα μέλη της οικογένειάς τους. Οπότε η ε, νόμιμη απόσπαση εργαζομένων στην Ευρώπη, έτσι όπως προτείνεται μέσα στις οδηγίες, θα καταστήσει αυτή τη δυνατότητα εντελώς αδύνατη. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Γιουγκέριος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σας για τη συζήτηση. Είναι πολύ χρήσιμο όλα αυτά τα στοιχεία για να οργανώσουμε και εμείς τις μελλοντικέ μας εργασίες για τούτη την πρόταση για την ισορροπία επαγγελματικού οικογενειακού βίου. Και θα ήθελα να μιλήσω για κάτι που αναφέρθηκε πιο πριν σε σχέση με τη σχέση της επίσημης και ανεπίσημης παροχής φροντίδας. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένας συνδετικός κρίκος στην ισορροπία οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Μιλήσατε για το ποσοστό των ατόμων που ε, δουλεύουν στην παροχή, στον τομέα της παροχής φροντίδας και είναι χαμηλόμιστοι και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν συνήθως άτομα να, δεν έχουν τα χρήματα συγγνώμη, για να προσλάβουν άτομα για να τους παράσχουν φροντίδα. Στην πρόταση Κομισιόν για την ε, παροχή φροντίδας αναφέρεται ότι ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα σε τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες άδεια το χρόνο. Αυτό δεν είναι αρκετό. Για τα άτομα που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις, όπου χρειάζεται ένα άτομο παροχής φροντίδας για ε, μακροχρόνια διαστήματα. Μιλήσατε για την επιλογή μη. Βεβαίως είναι και επιλογή το πώς θα αντιμετωπίσει κανείς, την, πώς θα απαντήσει στην κατάσταση που του προκύπτει. Αν έχει ένα παιδί ή ένα άτομο με αναπηρία ή έναν ηλικιωμένο στην οικογένειά του που χρήζει φροντίδας και ουσιαστικά βασίζεται στην παροχή του από αυτόν τον άτυπο φροντιστή. Το ερώτημα μου είναι, Αν μία οικογένεια με έναν συγγενή που υποφέρει ας πούμε από μία μόνιμη αναπηρία και χρειάζεται φροντίδα κατά τη διάρκεια των ημερών εργασία. Ε, κατάλαβα και αυτό που είπατε για τις ευέλικτες ώρες, ε, το ευέλικτο ωράριο. Αυτό να αποτελεί λύση όντω για πολλά προβλήματα, αλλά όχι για όλες τις περιπτώσεις όπου ο ε, εργαζόμενος ας πούμε έχει πολύ χαμηλό εισόδημα και κάποιος με ένα μόνιμο χρόνιο πρόβλημα υγείας βασίζεται σε αυτόν για να του παράσχει βοήθεια. Οπότε το ερώτημά μου είναι εμείς εδώ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα για να διασφαλίσουμε την ε, φτηνή ε, παροχή φροντίδας και τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών φροντίδας. Πέραν των πέντε ημερών δηλαδή της άδεια, ποια είναι τα επόμενα βήματα που μπορεί να υπάρξουν. Και αν μπορείτε, πείτε μας λίγο για τα κριτήρια της Βαρκελόνης και κατά πόσο αυτά μπορούν να βοηθήσουν αυτό το θέμα ένα ερώτημα είναι αυτό. Το άλλο ερώτημα είναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή επίσημα δεδομένα σε ό,τι αφορά την, το κόστος της επίσημης παροχής φροντίδας, δηλαδή έχουμε στοιχεία στατιστικά για να μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτά για τα άτομα με τις αναπηρίες, τα κρατημέλη ας πούμε και την παροχή φροντίδα σε αυτά. Έχουμε κάποια εσωτερική εικόνα για τη διαφορά της τιμής της, παροχής, της αξίας της παροχής φροντίδας και του μισθού που δίδεται στα κρατημέλη έτσι ώστε να έχουμε, πόσο μεγάλο είναι το, να έχουμε μια ιδέα για το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα ή το χάσμα. Έχουμε τα χαμηλά εισοδήματα, έχουμε τις πέντε ημέρες άδεια για τους άτυπους φροντιστές, νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα. Αλλά αν έχετε κάποια δεδομένα επίσημα, θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να μας τα δώσετε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Σιντνάνσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σλοβαγικά, οπότε παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές γιατί κάνανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ο καθένας τους. Το θέμα είναι σημαντικό και είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί εδώ και χρόνια. Πιο συγκεκριμένα ε, ασχολούμαι με οικογένειες που έχουν παιδιά με αναπηρίες. Και όπως ε, ακούστηκε πολύ συχνά εδώ, οι οικογένειες αυτές πραγματικά κινδυνεύουν από τη φτώχεια και πολύ συχνά αποδομούνται. Γιατί, Γιατί έχουν αυτό το παιδί με την αναπηρία, με το οποίο πρέπει να μείνει μόνη η μητέρα ε, να το φροντίζει, γιατί τα χρήματα για 24 ώρη φροντίδα όλο το μήνα είναι πάρα πολύ μεγάλα, πάρα πολλά. Οπότε όταν υπάρχουν οι υπηρεσίες εντάξει, αλλά υπάρχουν και κάποιες υπηρεσίες που θα έπρεπε να αναλάβουν οι αρχές, οι δημοτικές, οι κρατικές, αλλά δυστυχώς στη Σλοβακία αυτό δεν συμβαίνει και κάναμε μια έρευνα και είδαμε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες προσφέρουν μόνο το 30% των δήμων στη χώρα μου. Το 70% δεν προσφέρει τίποτα σε αυτούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι βάρος είναι το να φροντίζει κανείς παιδιά τα οποία έχουν αναπηρίες και αυτό βαραίνει ε, συνήθως τη μητέρα της οικογένειας και βέβαια στα πλαίσια αυτά προκύπτουν και δύο θέματα. Και μεγάλη χαρά θα σχολιάσω το εξή. Υπηρεσίε στήριξη της οικογένεια. Δηλαδή, θα πρέπει οι υπηρεσίε αυτές να μην εστιάζουν μόνο στο άτομο που χρειάζεται τη φροντίδα ή στο παιδί με την αναπηρία, αλλά σε ολόκληρη την οικογένεια. Για παράδειγμα, μπορεί στην οικογένεια το ένα παιδί να, είναι, ε, να έχει μια αναπηρία και το άλλο παιδί να μην έχει. Ε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, ε, και αυτό είναι η προσπάθεια στην Σλοβακία, είναι οι υπηρεσίε που στηρίζουν την οικογένεια να προσφέρονται και στο παιδί το οποίο έχει την υγεία του. Ε, στην περίπτωση που το, η μητέρα μένει στο σπίτι με το παιδί που έχει αναπηρία, θέλει κάποιον, για παράδειγμα, να της να το παιδί στο σχολείο το παιδί που πάει σχολείο. Άρα λοιπόν αυτές οι υπηρεσίες, η φροντίδα, ε, όταν πρέπει να καθαρίσουν το σπίτι του, όταν πρέπει να πάνε να ψωνίσουν. Χρειάζονται λοιπόν αυτή την επιπλέον βοήθεια και αυτή η βοήθεια προσφέρεται συνολικά στην οικογένεια, όχι μόνο στο άτομο που έχει την αναπηρία. Το δεύτερο, και είναι πολύ σημαντικό και αυτό, είναι ε, πώς μπορούν να αμείβονται αυτοί οι άνθρωποι που προσφέρουν φροντίδα, που είναι αυτές οι γυναίκες, που είναι πολύ άξιες που βοηθάνε και που χρειάζονται και πολλές ιατρικές ε, ε, γνώσεις. Για παράδειγμα, χρειάζονται κάποιες ε, λογοπαιδικές ε, γνώσεις, κάποιες φυσιο, γνώσεις φυσιοθεραπείας, γιατί κάνουν πολλές φορές θεραπεία αποκατάστασης και ένα σωρό άλλους δεξιότητες. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σπουδάσει μια ζωή και δεν ξέρουν τόσο πολλά αυτές οι γυναίκες. Χρειάζονται λοιπόν να αποκτήσουν αυτές τις ε, δεξιότητες, ε, να τις χρησιμοποιήσουν και εμείς θα πρέπει να τις αναγνωρίσουμε και να τις αντιμετωπίσουμε γιατί τη στιγμή που ε, ένας πατέρας ή μια μητέρα όταν αφού περάσει ένα χρόνο με την οικογένειά του και μετά πια δεν χρειάζεται να είναι συνέχεια εκεί θέλει να μπει στην αγορά εργασίας αυτές οι δεξιότητες που έχει αποκτήσει πρέπει να αναγνωρίζονται γιατί έχω γυναίκες που μου λένε έμεινα στο σπίτι με την οικογένειά μου 10 χρόνια δεν ξέρω τίποτα μα και βέβαια ξέρουν έχουν ειδικέ ε, γνώσεις οι οποίες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι οποίες θα πρέπει να ανταμείβονται με κάποιο τρόπο. Ξέρω πως το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά περίπλοκο, είναι πάρα πολλά τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε και με μεγάλη χαρά θα βρω μαζί σας κάποιες λύσεις για ερωτήματα γιατί θέλουμε πραγματικά να είναι πιο αξιοπρεπές το καθεστώς για τους ανθρώπους που φροντίζουν άλλους στην Ευρώπη. Ο κύριος Ροκφόρτ παρακαλώ. Okay. You didn't ask for the floor. Κύριε Ροσφόρ, δεν ζητήσατε το λόγο. Άρα είναι η κυρία Χάρκιν. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω όλους μας τους ομιλητές και πρέπει να σας πω ότι με αρκετό από αυτούς είμαι πολύ εξοικειωμένη γιατί είμαστε στην ομάδα που προσπαθεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ανθρώπων που φροντίζουν αλλά κάτι που ακούσαμε σήμερα και δεν το ακούμε συχνά στη Κοινοβουλή είναι το γεγονό πως και οι τέσσερις που κάνατε μία παρουσίαση είπατε πως συμφωνείτε πως η πρόταση αυτή είναι θετική. Ε, αυτό να το θεωρήσω βήμα προς σωστή κατεύθυνση και πιστεύω πως και εσείς πρέπει να γνωρίζετε πως η Επιτροπή μας και όλο το Κοινοβούλιο σε αρκετές περιπτώσεις μέσω ψηφισμάτων κτλ. έχει ψηφίσει και έχει ζητήσει να περάσει να περάσουν πολλά από αυτά τα στοιχεία του πακέτου, γιατί πολύ συχνά μιλάμε για το δημοκρατικό έλλειμμα μεταξύ των όσων κάνουμε εμείς εδώ και όσων συμβαίνουν στην πραγματική ζωή, αλλά νομίζω ότι για εδώ μπορούμε να πούμε πως ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Οπότε Τώρα λοιπόν που σας επένεσα και μας επένεσα, πρέπει να δούμε και τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Και έχω αρκετέ ερωτήσεις και ένα σχόλιο. Τι είπε οι Eurocarers. Πολύ συχνά ο κόσμος δεν έχει επιλογή. Γι' αυτό λοιπόν, αν δούμε όσους ε, είναι άτομα που φροντίζουν την οικογένειά τους με άτυπο τρόπο, θα δείτε πως είναι ένας βασικός πυλώνας που στηρίζει ε, τα συστήματα δημόσιας υγείας και περίθαλψης στην Ευρώπη, τα οποία θα κατέρεαν γιατί ε, δεν μπορούμε να βρούμε αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι επίσημα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Χρειάζεται και αυτό το ανεπίσημο συστατικό στοιχείο που έχει να κάνει με το πώς είναι στημένη η κοινωνία μας και ποιες είναι οι δημογραφικές πιέσεις που καλύπτουμε. Όλοι ζούμε περισσότερο, αυτό είναι θετικό. Όμως, Γι' αυτό έχουμε και την πρόταση τούτη που είναι τόσο σημαντική. Οι ερωτήσεις λοιπόν που έχω να κάνω είναι οι εξής. Καταρχήν, αρκετοί συνάδελφοι μίλησαν για την ανάγκη του να παρατείνουμε τη μία εβδομάδα και ξέρω πως αρκετά κράτη έχουν διαφορετικά συστήματα. Στην Ιρλανδία εμείς έχουμε κάτι ε, πολύ ε, ευρύτερο για αυτή την δυνατότητα άδεια. Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί στις χώρες που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και να δούμε αν μπορούμε να το εφαρμόσουμε και αλλού. Και ίσως κάπου μπορούμε να κάνουμε και μια βελτίωση της πρότασης. Θεωρείτε πως είναι πολύ φιλόδοξο αυτό, γιατί όλοι είπαμε ότι χρειάζεται. Μήπως είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι για το πόσο άδεια χρειάζεται. Δεύτερον, μιλήσατε για ευελιξία. Και η συνάδελφος από την Πολωνία μίλησε για, τη, για το εξατομικευμένο δικαίωμα για γονική άδεια και πώς πρέπει να πείσουμε τους εργοδότες και να τους προωθήσουμε, να τους σπρώξουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ρωτώ όλους, πιστεύετε πως πρόταση αυτή μπορεί να έχει παρόμοιο αποτέλεσμα, τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε τη δυνατότητα αυτή και να είναι θετική η έκβαση. Επίσης, δεν θα πρέπει να ντραπούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να έχουμε και εκεί ευελιξία. Ευελιξία και παράλληλα μικρομεσαίες να μην μας πούνε πάλι μα αν τα περάσουμε όλα αυτά θα χάσουμε τη δουλειά μας. Γιατί εντάξει, υπάρχουν ορισμένε φορέ δύσκολα ερωτήματα στη ζωή, αλλά με το να κλείνει τα μάτια κανεί δεν τα λύνει. Εμεί σήμερα μιλήσαμε πολύ για το θέμα του φίλου. Έχετε στοιχεία? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς, φροντίζουν είναι οι γυναίκες, πώς οι άνδρες. Θα έλεγα ότι στην Ιρλανδία είναι 60-40, γιατί όλο και περισσότεροι άντρε αναλαμβάνουν το ρόλο αυτό. Αλλά δεν ξέρω Ίσως σε άλλα κράτη τα πράγματα να είναι κάπως διαφορετικά. Έχετε στοιχεία? Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ. Καλό είναι που το συζητάμε το θέμα αυτό. Και έχουμε και την πρόταση για την ε, ισορροπία επαγγελματικού οικογενειακού βίου στο τραπέζι, οπότε μιλάμε για πράγματα της πραγματικής ζωής. Και θα ε, σας παραπέμψω και εγώ στο σλοβακικό παράδειγμα. Ήταν πραγματικά πολύ ακριβές. Και πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο για την ε, επαγγελματική παροχή φροντίδας από τους ε, φροντιστές, για την τυποποίηση των, ε, του σχετικού επαγγέλματος, αλλά και, τον, και τη δυνατότητα ανέλυξης στην επαγγελματική ιεραρχία στον τομέα αυτό. Είναι σημαντικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό να γίνουν αντίστοιχε πράξει. Πάμε στο ερώτημά μου. Οι ε, παροχή φροντίδα παίρνουν 50% ή παραπάνω ε, αυτών, αυτών που ουσιαστικά δίνουν στο άτομο για να παράσχει την ε, φροντίδα. Υπάρχει τρόπος να ρυθμίσουμε λίγο τις εταιρείες οι οποίες παρέχουν αυτούς τους φροντιστές στις διάφορες οικογένειες που τους χρειάζονται. Ο κύριος Μάρτιν. Ο κύριος Μαχτά, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, όλους τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά πραγματικά λυπούμε. Μάλλον θα χαλάσω το κλίμα. Διότι πρέπει όλοι να αποδεχτούμε τις αντιφάσεις που μας αφορούν και εδώ υπάρχει μία που νομίζω ότι είναι θερμοφανή. Ε, όλοι θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των οικογενειών και των φροντιστών. Πολλέ φορέ είναι γυναίκε, πολλέ φορέ είναι άνθρωποι που εργάζονται ε, σε κάποιο κατάστημα, ε, σε κάποιο σε κάποια γεωργική εκμετάλλευση. Τέλος πάντων, πρέπει να σκεφτούμε τι είδου κοινωνία θέλουμε να φτιάξουμε. Εντάξει, είναι καλή αρχή που προτείνει η οδηγία, συμφωνώ όμως υπόθηκαν, αλλά Πρέπει να σκεφτούμε για την κοινωνία μας τι μοντέλο θέλουμε πρώτα απ' όλα. Αυτά που προτείνετε, αυτά που λέτε και λέω και εγώ, είναι τελείως τους αντίποδες, αντιδιαμετρικά αντίθετα με τους δημοσιονομικούς προσανατολισμούς της Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τέλος πάντων μάλλον καλύτερα του Συμβουλίου, γιατί μην είναι αυτά που το μαθα, τα κράτη είναι, είναι να μειώσουμε προς τα κάτω τις ε, δαπάνες. Πώς θα πληρώσουμε όλο λιγότερα, όσο δυνατόν λιγότερα οι κοινωνικέ δαπάνε ονομάζονται κοινωνικό βάρο. Σημαίνει ότι του βαραίνουν να τα μειώσουν. Άρα εδώ υπάρχει μια ε, εκ των πραγμάτων αντίφαση. Δηλαδή η οδηγία είναι πολύ ωραία, μπορεί να εμποδίσει τους εργαζομένου το, της Ευρώπη, Ευρώπης να έρθουν προ τα δυτικά να περιθάλψουν ε, αρρώστου ή αυτού που έχουν ανάγκη. Και θα βοηθήσει κακοπληρωμένου εργαζομένου τη Δυτική Ευρώπη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και οι εργαζόμενοι τη Ανατολική Ευρώπη έχουν οικογένειε και πρέπει και αυτοί να προστατευτούν. Ε, εδώ λοιπόν, τι θα κάνουμε, μια και έχουμε ψηφίσει τον προπολογισμό, θα φανούμε γενναιόδοροι και θα πούμε δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτό. Εκατομμύρια άτομα σήμερα δεν λαμβάνονται υπόψη, του έχουν εγκαταλείψει στην τύχη του, δεν αυτή η σύγχρονη κοινωνία που θέλουμε και μετά Διερωτώ με, το Συμβούλιο θα δεχτεί αυτά που λέμε τώρα εδώ να ισχύσουν ας πούμε και για τον ελληνικό λαό, ενώ τους γδίσαμε, τους γδίσαμε τελείως, τους εξαπατήσαμε και συνεχίζουμε να τους εξαπατούμε. Και τους παίρνουμε ό,τι τους έχει μείνει. Τους έχει μείνει ίσως ένα ρούχο, ε, ένα πουκάμισο και ένα παντελόνι με το ζόρι, ένα βρακί. Ε, τι υποκρισία είναι αυτή. Ε, εδώ πρέπει να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Το ερώτημα είναι ποιο πληρώνει. Ποιο. Δεν απευθύνομαι επιθετικά σε εσά, διότι εκπροσωπείτε και του γεωργού κάποιε φορέ. Ε, ε, αλλά Κάποιοι έρχονται εδώ να μας πούνε ε, πληρώνουμε πολλά βάρη, πολλούς φόρους. Οι πολυεθνικές πληρώνουν πολύ λιγότερους φόρους από εσά και από εμένα. Τους κάνουν δωράκια. Ε, δωράκια που κοστίζουν όμως έχουν βάρος ε, το αντίστοιχο σε χρυσό. Εδώ λοιπόν πρέπει να αποδεχτούμε ή τουλάχιστον να δούμε κατάματα της, ε, κατάφατσα της αντιφάσης μας. Ε, Στι διάφορε χώρε μα, στη δική μου τη χώρα, τη Γαλλία, ο πρόεδρο που μόλι κέρδισε τι εκλογέ δεν ήταν ο χειρότερο, αλλά είναι ένα υποψήφιο ο οποίο υποσχέθηκε στου Γάλλου τη μείωση των φόρων. Το καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό. Στο κεφάλι των ανθρώπων θα σημαίνει ότι θα μειώνονται μεν οι φόροι, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι οι φόροι είναι το κοινωνικό μα μοντέλο. Αυτό στηρίζει το κοινωνικό μα πρότυπο. Αυτό επιτρέπει να ζούμε όπω ζούμε. Εάν μειώνουμε διαρκώ του φόρου, διαρκώ τα βάρη και τα άχθη όπω ονομάζονται, ποιο θα πληρώνει. Ποιο θα πληρώνει. Το ερώτημα λοιπόν είναι, οι Έλληνε φίλοι και συνάδελφοι θα υποφεληθούν από αυτό το νέο πλεονέκτημα, αυτό το νέο προνόμιο. Είμαι βέβαιο πω όχι. Είμαι βέβαιο πω θα πούμε, Α, όχι, όχι εσεί, πρώτα θα πληρώσετε το χρέο και μετά βλέπουμε. Με συγχωρείτε, αλλά ήθελα λίγο να βάλω και τι φωνέ και να τα ψάλω σε όσου πρέπει να τα ακούσουν, γιατί από τη μια υπάρχουν πολλέ καλέ προθέσει, από την άλλη όμω υπάρχει και μια υποκρισία. Υπάρχει ο κόσμο τη κοινωνία των πολιτών, ε, των συλλόγων, σα λένε τι ωραίοι που είστε, τι καλοί, τι φανταστικέ ιδέε. Μ' άρεσαν πάρα πολύ ωραία αυτά που είπατε, ήταν υπέροχα. Καλύτερη ζωή για όλε τι οικογένειε χωρί εξαίρεση. Για τα 28 κρατημέλη, σοβαρά. Ε, Εμεί πρέπει να κάνουμε τη σωστή επιλογή. Από κοινού. Αυτό θα παιχτεί το 2019. Thank you. Mr. Hetman. Thank you, Madam Chair. Please. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πολωνικά, αν μου επιτρέπετε, οπότε φορέστε τα κωδικά σας, παρακαλώ. Oczywiście, poza panią profesor. Ε, ε, Szanowni Państwo. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, και εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, παρουσιάσεις σας, για όλα τα στοιχεία που μας ε, δώσατε. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες και εμπλουτίζουν τη συζήτηση που θα κάνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είμαι σίγουρος ότι σχεδόν όλοι ε, θεωρούμε ότι όλες οι ιδέες που μας παρουσιάσατε είναι πάρα πολύ καλές και είναι πολύ καλές συστάσεις σας. Και είναι πολύ θετικές οι απόψεις, ακόμα και ε, όταν μιλούμε για τους εργοδότες, γιατί ε, έχω, το έχω συζητήσει και εγώ το θέμα αυτό με ενώσεις εργοδοτών από την ε, Πολωνία και συμφωνούν απολύτως με την ιδέα που προτείνεται. Βεβαίω θα παρακολουθήσουν στενά το πώ θα εξελιχθεί. Ε, περνάμε τώρα στι λεπτομέρειε. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το θέμα αυτό ένα θέμα που πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ γιατί η, ιδέα της ισορροπίας της ε, εργασιακής και της οικογενειακής ζωής δεν θα πρέπει να καθιστά αδύνατο να δούμε τις λεπτομέρειες που την αποτελούν και μιλώ ως νέος πατέρας γιατί όταν μιλούμε για γονική άδεια, όταν μιλούμε για αυτή την, περίπτωση, αυτή την περίοδο όπου και η μητέρα και ο πατέρας ε, μπορούν να φροντίσουν το μωρό τους μετά την ε, γέννησή του, σκέφτομαι ο στόχος ακριβώς ποιος είναι. Να, φροντίσει το, να φροντίσουμε το παιδί, να το στηρίξουμε αυτή τη στιγμή γεννήθηκε. Η στήριξη, η φροντίδα που μπορεί να δοθεί από τους γονείς του είναι ο στόχος που βεβαίω αυτό ε, κάνει πάρα πολύ καλή τη ζωή του νεογέννητου ή ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι πατέρες θα φροντίζουν τα παιδιά τους. Γιατί νομίζω ότι ε, είναι σαφές και οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε μαζί μου, κάποιοι πατέρες δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα στήριξης για τα παιδιά τους. Και, όταν, και αυτή η περίοδος όπου ένας γονιός μπορεί να φροντίσει το παιδί του, ουσιαστικά χάνεται. Άρα αυτό υπονομεύει την ευημερία του μωρού. Το αντικείμενο λοιπόν της αναλυσής μας εδώ θα πρέπει να είναι το παιδί και η ευημερία του παιδιού, όχι μόνο του πατέρα και της μητέρας. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι όταν ε, μελετούμε τα θέματα αυτά πρέπει να τα μελετούμε εις βάθος. Και το ερώτημα είναι πώς αυξάνουμε την ευαισθητοποίηση και των εργοδοτών. Γιατί είμαι πεπισμένος, γιατί ξέρω εργοδότες που χωρίς ε, να τους το επιβάλλει ο νόμος, χωρίς κανόνες, έχουν εισαγάγει ευέλικτες συνθήκες εργασίας, γιατί ξέρουν ότι αυτό αυξάνει την ποιότητα ε, της εργασίας στην εταιρεία τους. Και το πιο σημαντικό στοιχείο εδώ είναι να αυξήσουμε την ε, παιδεία, την εκπαίδευση των, εργαζομε... των ε, εργοδοτών. Γιατί αν καταλάβουν ότι όντως είναι ε, ωφέλιμο για την εταιρεία τους, είναι πολύ πιο πιθανό να εισαγάγουν τέτοιες ρυθμίσεις υποστήριξης των γονιών που δουλεύουν στην εταιρεία τους. Πολύ σημαντική λοιπόν η συζήτηση αυτή για τους φροντιστές, για τους φροντιστές που, φροντίζουν ε, άτομα με αναπηρία, ε, ηλικιωμένους. Σε πολλές χώρες η θεσμική στήριξη είναι πολύ χαμηλή, κυρίως για τους ηλικιωμένους. Οπότε αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ θετική. Γενικώ λοιπόν θέλω να πω ότι η δουλειά μας εδώ είναι απλή. Πρέπει να αναλύσουμε τις νομικές συνέπειες, το νομικό αντίκτυπο στα κρατη Πρέπει να αξιολογήσουμε τα οικονομικά, κοινωνικά, τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο και αν όντως όλα αυτά είναι καλά, τότε μπορούμε όντως να συμφωνήσουμε. Δύο έχω ακόμη στον καταλογό μου για να πάρουν το λόγο και μετά θα δώσουμε το λόγο στους ε, προσκεκλημένους μας, δυστυχώς λίγο χρόνο έχουμε, ε, για να απαντήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά ο Γάλλος συνάδελφος με οδηγεί στο να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου. Εγώ ανήκω σε μια πολιτική ομάδα η οποία δεν θέλει να είμαστε κατά των κοινωνικών ε, μέτρων στην οικονομία, γιατί διαφορετικά θα κατεδικαστούμε σε μια κοινωνική ε, σε ένα κοινωνικό μαρασμό γιατί ξέρετε πως όταν δημιουργούμε θέσεις εργασίας μέσω της ανάπτυξης της οικονομίας, τότε ναι μπορούμε να πληρώνουμε και τις κοινωνικές παροχές. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας και νομίζω αρκετοί το είπαν και τους ευχαριστώ οι παρουσιαστές πως η γενικότερη βοήθεια που μπορεί να προσταφρεθεί από τους από τα μέλη της οικογένειας και από τους γείτονες είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι μπορεί να κάνουμε σε θεσμικό επίπεδο μέσω των αρχών. Οπότε θα πρέπει να το διατηρήσουμε γιατί ξέρετε οι οικογένειες είναι η πρώτη πηγή βοήθειας και θα πρέπει αυτό να αναγνωρίζετε. γιατί για πάρα πολλά χρόνια ήταν κάτι το αόρατο και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αναγνωρίζετε και να φαίνεται. Δυστυχώς όμως και δεν θέλω να είμαι κοινικός, μην νομίζω ότι κάνω αυτό το λάθος, αλλά όταν βοηθάνε οι οικογένειε είναι πολύ πιο φθηνό από το να το κάνει το κράτος. Οπότε ας βοηθήσουμε τις οικογένειε να βοηθούν και με τον τρόπο αυτό είναι θα είναι επιτυχημένο το κοινό μας μοντέλο, γιατί και σε ψυχολογικό επίπεδο είναι προτιμητικό για το άτομο που χρειάζεται βοήθεια και θα είναι και θετικός ο οικονομικός αντίκτυπος. Από τις μελέτες που έκανα στο παρελθόν είχα δει πως συγκεκριμένα για όσους φροντίζουν και δεν ξέρω αν οι εμπειρογνώμονες θα συμφωνήσουν, τουλάχιστον στη Γαλλία έτσι ήταν, είχαμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δεν ήθελε ας πούμε αμοιβή, αλλά ανησυχούσε πάρα πολύ επειδή έχανε συνταξιδοτικά δικαιώματα, επειδή δεν δούλευε γιατί φρόντιζε κάποιον στην οικογένειά του. Οπότε μία από τις προτεραιότητες θα είναι να δούμε τι γίνεται, όταν κάποιος λοιπόν φροντίζει ένα μέλος οικογένειας να μην χάνει δικαιώματα συνταξιοδοτικά και να μπορεί να συνεχεί να σωρεύει δικαιώματα διαφορετικά Κάποιοι θα λένε, ξέρετε, εγώ μπορώ να διακόψω την επαγγελματικό μου βίο για να βοηθήσω, αλλά δεν το κάνω, γιατί καταλαβαίνετε τι θα συμβεί. Θα πληρώσω διπλά ούτε μισθό θα παίρνω σήμερα και όταν αύριο θα είμαι συνταξιούχος η σύνταξή μου θα είναι χαμηλότερη γιατί δεν θα έχω πληρώσει αρκετές εισφορές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα διπλό πρόβλημα. Χρειαζόμαστε λοιπόν να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς και αυτό που γινόταν παλιά οι άνθρωποι έβγαιναν στη σύνταξη στα 60-61 και τότε μπορούσαν να βοηθήσουν παρόλο που δεν εργαζόντουσαν και έπαιρναν σύνταξη. Επειδή όμω τώρα βγαίνουμε στη σύνταξη αργότερα, υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που 60, 61, 62 ετών που σήμερα εργάζονται. Δεν είναι πλέον συνταξιούχοι, οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτούς. Και πήρα το λόγο γιατί ήθελα να κλείσω με το εξή. Στη χώρα μου, τη Γαλλία, νομίζω ότι στο θέμα αυτό προχωράμε. Και είναι καλό να προχωρήσουμε και στην Ευρώπη. Δεν θέλω να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες. Να πω μόνο πως τα άτομα τα οποία είναι εξαρτημένα έχουν δικαίωμα σε βοήθεια, η οποία συνήθως είναι ανεπαρκής σε δημόσια βοήθεια, κρατική βοήθεια. Και σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να είμαστε μισθοδοτούμενος όταν φροντίζουμε την οικογένειά μας, πώς πως ε, λαμβάνοντας ως μισθό το επίδομα που πληρώνει στην οικογένεια το κράτος. Έχουμε ένα είδος ανταλλαγής ας πούμε, έτσι ώστε υπολογίζουν την οικογενειακή, το, το οικογενειακό επίδομα που θα πλήρωνε το κράτος σε κάποιον άλλο και το δίνει στον άνθρωπο από την οικογένεια που φροντίζει. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κούνεβα, τελευταία ομιλήτρια. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ σήμερα για την συζήτηση αυτή που κάνουμε. Χαίρομαι γιατί ακούω όλες τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει στην έκτηση που κάναμε πριν ένα χρόνο για το οικιακό προσωπικό, αλλά και σε άλλα ψηφίσματα των δύο επιτροπών να προτείνουμε εδώ από τους που προτείναμε από τους επιλογνώμενους που συζητήσαμε εδώ. Είχαμε συνεργαστεί μαζί τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω πως επειδή το θέμα της ισορροπίας οικογενειακής και εργασιακής ζωής επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τη δουλειά μας με συνεργασία των δύο επιτροπών της Επιτροπής Επασχόλησης και της Επιτροπής Γυναικών. Εγώ ήμουν η συγκίτρια την Επιτροπή ε, γυναικών, αλλά η δουλειά μου δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς τη συμμετοχή της Επιτροπής Απασχόλησης. Το ίδιο θα είχε και την Επιτροπή Απασχόλησης. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, επηρεάζει πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων και αν δεν έχουμε την μεγαλύτερη συνεργασία δεν θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, να ακούσουμε και ένα σύντομο σχόλιο, ίσως, από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Δύο εκπρόσωποι εδώ υπάρχετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένας από εσά μπορεί να πάρει το λόγο για να αφήσουμε και λίγο χρόνο στους εμπειρογνώμονες να απαντήσουν. Ευχαριστώ. Μανουέλα Γκέλινγκ ονομάζομαι από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για, για τα πολύ θετικά επικοδομητικά σχόλια που ακούσαμε σήμερα. Όντω, η ισορροπία ε, για την. Η πρόταση, μάλλον και το πακέτο που προτείνει η Κομισιόν για την ισορροπία επαγγελματικού και οικογενειακού βίου προσπαθεί να καλύψει τι ε, προκλήσει ό,τι αφορά την απασχόληση και την ανεργία, γιατί ε, πολλέ γυναίκε υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασία και την, το θέμα της ηλικία, γιατί οι γυναίκε που δεν έχουν υπάρξει πολύ, για πολύ καιρό στην αγορά εργασία αντιμετωπίζουν την απειλή τη φτώχεια και το γεγονό ότι βεβαίω η κοινωνία αλλάζει. Η, η πρωτοβουλία λοιπόν βλέπει και τις, ε, όλες τις δέσμες δικαιωμάτων που υπάρχουν στην πρόταση οδηγία, αλλά μελετά και άλλες πολιτικές χρηματοδοτικών μέσων. Ας πούμε δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για την μακροπρόθεσμη φροντίδα για τα, για τα παιδιά, αλλά είδαμε ότι πρέπει να υπάρξει τέτοια δυνατότητα χρηματοδότησης ή καλύτερη εποπτεία των δεδομένων. Το είπατε πολύ το θέμα των δεδομένων και επίσης σε κάποια benchmarks στην, σε ό,τι αφορά τη μακρόχρονη φροντίδα των παιδιών. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο τώρα. Πολύ σημαντικός τομέας όπου θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ε, έμφαση στην ισορροπία επαγγελματικού οικογενειακού βίου και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει σε έναν βαθμό τα προηγούμενα χρόνια. Θα ήθελα να μιλήσω για κάποια σχόλια που έγιναν. Η ισορροπία οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, έτσι όπως προτείνεται, μελετά καταρχάς τη δημιουργία ε, θεμητών και δίκαιων συνθήκων εργασίας για άντρες και γυναίκες στην αγορά εργασία, ε, για την αντιμετώπιση της ισότητας των φύλων, αλλά και για τα ωφέλη ό,τι αφορά την κοινωνία, την οικονομία και, το, και τα κράτη. Έγινε και ένα, ετέθη ένα ερώτημα για το κόστος, ή το σύνολο της πρότασης. Μιλά για το ότι τα ωφέλη ε, θα είναι περισσότερα από το κόστος. Και σίγουρα θα υπάρχουν ε, ε, και για τους άντρες και για τις γυναίκες ωφέλη, αλλά και για τις οικονομίες και για τα κράτη. Η συμμετοχή τώρα των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι επίσης το σημείο κλειδί και Γι' αυτό όταν ε, βλέπουμε το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες μέρες άδεια, η φιλοσοφία εδώ λέει ότι μελετούμε το ότι αν μείνει κανείς εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε έχει λιγότερες ευκαιρίες να απασχοληθεί και να προχωρήσει στην καριέρα του. Και γι' αυτό έχουμε, η πρόταση έχει γίνει για πέντε μέρε μόνο και όχι περισσότερο. Ξέρουμε ότι τα, κάποια κρατημέλη έχουν περισσότερε ημέρε. άδεια. Αυτή είναι μια πρόταση οδηγία του ή άλλου, που θέτει ελάχιστε ε, προϋποθέσεις. Τα κρατημέλη φυσικά έχουν πάντα το ελεύθερο να τι ξεπεράσουν. Επίση, είδαμε το είδο των ατόμων που, μπορούν να, που δικαιούνται αυτή την άδεια για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει σωστό. ε, διαμερισμός μεταξύ αντρών και γυναικών και νομίζω ότι αυτό έχει αναφερθεί ρητά στην οδηγία, στην πρόταση, ε, Για τη συγκρισιμότητα τώρα των δεδομένων, για την μακροχρόνια φροντίδα. Όντως, δεν έχουμε συγκρίσιμα δεδομένα στη φάση αυτή. Αλλά έχουμε ξεκινήσει μία μελέτη για να δούμε τη μεθοδολογία που θα μας επέτρεπε να έχουμε συγκρίσιμα δεδομένα για την μακροχρόνια φροντίδα. Τώρα, οι μέρες ε, άδεια που έχουμε προτείνει δεν είναι υποχρεωτικές, είναι επιλογή του καθενός αν θα τις πάρει όχι. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα την οπτική το πώς αυτό επηρεάζει το παιδί, οι μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά εποφελούνται από τη συμβολή και των δύο γονιών, οπότε η μαθησιακή τους εξέλιξη θα είναι πολύ καλύτερη αν και οι πατέρες και οι μητέρες εμπλέκονται στην ανάπτυξη του παιδιού. Αυτά νομίζω. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε. Κύριε Ηγεμόνος σύντομε παρατηρήσεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ευχαριστώ θερμά για τις ερωτήσει. Πέντε μέρες. Θα θέλαμε περισσότερες. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν χώρε που δεν έχουν τίποτα. Οπότε ίσως να είναι θέμα επιφυλακτικότητας λόγω της εμπειρία που είχαμε και με την άδεια μητρότητας. Κάτι είναι για αρχή οι πέντε μέρε. Εάν δεν κάνω λάθο, τα συνοδευτικά έγγραφα της Επιτροπής εξηγούν ότι η πενταήμερη άδεια είναι το ίδιο ε, με το κόστος ε, των συστηματικών αποσυρών. Δηλαδή 0, κάτι δεν θα κοστίσει τίποτα εάν λάβουμε υπόψη τις συστηματικές αποσύσεις, ε, Για την κοινωνική διάσταση και την υγειονομική σε συνδυασμό και πάλι η ισορροπία επαγγελματικού οικογενειακού βίου ω ε, έγγραφο κείμενο είναι μέρο ενό μεγαλύτερου παζλ, μια συνολικότερη εικόνα. Πρέπει να δούμε και την τελική διακοπή του πυλώνα πριν αποφανθούμε και πολλά λέγονται στην Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ για να βρουν πώς θα μπορέσουν όλοι να εντοπιστούν ε, στο βασικό τομέα υγείας, τι θα γίνει με τους φροντιστές και πώς διαφορετικές καταστάσεις θα εξεταστούν παράλληλα. Είναι σε εξέλιξη όλο αυτό. Η προσέγγιση από τη σκοπιά των οικογενειών, πολύ καλή προοπτική και μου δίνει την ευκαιρία να σας αναφέρω και ένα άλλο είδος φροντιστών που είναι τελείως αόρατοι. Οι νέοι φροντιστές κάτω των 18 που δεν καταγράφονται πουθενά που δείχνει ότι μπορεί δύο παιδιά να έχουν ευθύνες στην Ευρώπη και μάλιστα έχει γίνει μια μελέτη που τους καταγράφει ένα τάξη σχολείου. Και είναι 5-6 παιδιά σε κάθε τάξη αυτά. Ε, εδώ λοιπόν Έχουμε μια πλατφόρμα με online εκπαίδευση για τους φροντιστές για να μπορούν να καλύψουν καθημερινές τους ανάγκες. Αλλά επίσης κάτι άλλο μας ενδιαφέρει είναι οι δεξιότητες που αναπτύσσει κανείς κατά την άσκηση των καθηκόντων της φροντίδας να μπορούν να πιστοποιηθούν. Στην Ευρώπη υπάρχει ακόμη πολύ επιφυλακτικότητα ως προς αυτό, όμως υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ιδίως από τους πολιτικούς ευθύνοντες. Θα θέλαμε λοιπόν να το διερευνήσουμε στο μέλλον. Αξιολόγηση των υπηρεσιών φροντιστών. Συνεργαζόμαστε πολύ με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση για την ε, κατάρτιση. Ελπίζουμε δικτών για τη μακροπρόθεσμη φροντίδα, οι οποίοι θα προβλέπουν και μέτρα υποστήριξη για του φροντιστέ, πρόσβαση και ποιότητα, οπότε και αυτό σε εξέλιξη. Η ανάλυση ανά το φύλλο και βάσει των αριθμών που έχουμε στα χέρια μα, 75% των φροντιστών στη γυναίκα, ε, στην Ευρώπη είναι γυναίκα. Είναι γυναίκες. ανάλογα με τις χώρες. Ε, για να το πω απλούστερα, στις σκανδιναβικές ή δυτικές χώρες είναι, 60, είναι 45-65%, στις μεσογειακές χώρες είναι καταστροφική πλειοψηφία γυναίκες. Πώς να πείσουμε τις εταιρείε. Σωστό, αλλά είναι τεράστιο το ε, όφελος. Τελευταία κουβέντα το υπόσχομαι. Ε, Υπάρχει εκστρατεία του Employers for Carers, ε, η πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, που ξεκίνησε υπηρεσία συμβουλευτική προ του εργοδότε και έχει απευθυνθεί σε μεγάλε εταιρείε όπω η British Telecom, οι οποίοι συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει τεράστιο θετικό αντίκτυπο για τι επιδόσει των εργαζομένων. Οπότε υπάρχει πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να δράσω για δύο πράγματα. Μιλήσαμε για το κόστος και το ποιος θα το αναλάβει. Εγώ θα μιλήσω λοιπόν για το κοινωνικό κόστος, γιατί στην Ευρώπη και στο Βέλγιο, αν θέλουμε το κοινωνικό καθεστώς των γυναικών που είναι στη γεωργία να το βελτιώσουμε, θα πρέπει να συνεισφέρουν οι ίδιες. Μέσω μιας κοινωνικής ασφάλισης, ε, έτσι ώστε το καθεστώς που θα τους προσφέρουμε να είναι καλύτερο, οπότε αν πληρώνουν κοινωνικές εισφορές θα πρέπει το καθεστώς αυτό να είναι κάτι το οποίο θα είναι όλο και καλύτερο. Και για την περίθαλψη και τη φροντίδα της οικογένεια υπάρχουν συστήματα τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν. Στο Βέλγιο για παράδειγμα έχουμε εισάγει εδώ και καιρό αυτές τις επιταγές, voucher δηλαδή, όπου οι οικογένειες πληρώνουν για φροντίδα στο σπίτι ε, ε, σε με μειωμένη τιμή και αυτό σε σχέση με το εισόδημα, δηλαδή έχει εισοδηματικά κριτήρια κτλ. Δηλαδή μεταξύ 5 και 9 ευρώ την ώρα και τα υπόλοιπα τα πληρώνει το κράτος. Αλλά θα πρέπει να καταλάβετε πως τα συστήματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να έχουμε πολλή δουλειά στη μαύρη και να είναι περισσότερα τα άτομα τα οποία δεν είναι δραστήρια στον αγορά εργασία και παρόλα αυτά που πληρώνουν φόρους ε, και πληρώνουν και εισφορέ. Οπότε θα πρέπει να συνδυάσουμε τις οικογενειακές παροχές και τα ε, προνοιακά επιδόματα με κάποιο είδους κοινωνική εισφορά έτσι ώστε να βρούμε μια ισορροπία. Και αυτά σε σχέση με την παρατήρηση που κάνατε για το ενδεχόμενο κόστος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κατόφσκα. Εγώ θεωρώ πως η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ σωστή και νομίζω θα μας ευιστοποιήσει καλύτερα στην ανάγκη για πραγματικά στοιχεία. Στοιχεία γιατί ανάγκες έχουμε σε τέτοιου είδους φροντίδα, γιατί στις χώρες μας είναι κατακαιρματισμένες οι υπηρεσίες, οπότε χρειαζόμαστε επίσημα στοιχεία γιατί συνήθως αυτά τα προσφέρει το Υπουργείο το σχετικό που δίνει τα στοιχεία για τις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας, αλλά χρειαζόμαστε και στατιστικά δεδομένα από στατιστικές έρευνες για να δούμε τι γίνεται με αυτές τις δράσεις που ε, έχουν σχέση με την φροντίδα στην οικογένεια. Οπότε θα πρέπει οι στατιστικές υπηρεσίες να κάνουν κάποιο είδους έρευνες και στα ιστακτικές ε, δημοσκοπήσεις που κάνουν να ρωτάνε να κάνουν τέτοιου είδου ερωτήσει. Δηλαδή, μιλάμε για την. Ε, ε, ε, Συνήθω στέλνουν ερωτήσει για την οικονομική δραστηριότητα, αλλά όχι για την. για την φροντίδα που προσφέρουμε και αυτά θα μπορούσαν να κάνουν στα πλαίσια της απογραφής που γίνεται κάθε δεκαετία. Θα ήθελα να απαντήσω και στην ερώτησή σας για τις οικογένειες με παιδιά με αναπηρίες, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και σημαντικό θύμα. Μπορώ να σας πω τι γίνεται στην Πολωνία. Κατά τη γνώμη μου, εδώ υπάρχει ένας κατακαιρματισμός και σε υπουργικό επίπεδο, γιατί στο Υπουργείο Υγείας έχουν κάποιες πληροφορίες, αλλά παράλληλα έχουν πληροφορίες και στο Υπουργείο Οικογένειας, Κοινωνικής Πολιτικής και Εργασίας. Και παράλληλα έχουν και αντίστοιχα στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω πως εδώ υπάρχει ο ακτιβισμός των γονέων των παιδιών αυτών που θα πρέπει να δημιουργήσουν κάποιο είδους ίδρυμα ή ένωση έτσι ώστε και τα δικά τους και οι δικές τους ανάγκες να ακούγονται. Γιατί δεν υπάρχει πραγματική κρατική δράση που να απευθύνεται στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Και το τελευταίο μου σχόλιο έχει να κάνει με τις συνέπειες στα ατομικά δικαιώματα για τη γονική άδεια. Νομίζω πως εμείς θεωρούμε πως πρέπει να υπάρχει χρονική επένδυση και των δύο γονέων στην οικογενειακή ζωή και στα παιδιά και θα πρέπει να βασιστούμε στις εμπειρικές μας αποδείξεις που αποδεικνύουν πως όσο περισσότερο χρόνο περνάνε οι πατεράδες με τα παιδιά, τόσο πιο θετικά είναι τα αποτελέσματα και στον τρόπο που αναπτύσσουν τα παιδιά και στον τρόπο που εργάζεται η γυναίκα και στον τρόπο που μπορεί κανείς να συμφιλιώσει τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Και μια τελευταία πρόταση είναι μια συζήτηση με τις ενώσεις εργοδοτών ε, όταν ε, εισήχθη η εξάμεινη γονική άδεια στην Πολωνία και δεν ήταν οι εργοδότες κατά αυτής της διάταξης. Οπότε δεν είχαμε αντίδραση από τους εργοδότες. Αυτό διαπιστώσαμε πριν από δύο χρόνια, όταν συζητούσαμε το θέμα μαζί τους είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο γιατί βοηθά να αλλάξουμε τον τρόπο που κατανοούν και οι εργοδότες τα θέματα αυτά. Δεν θα πρέπει να μελήσουμε λοιπόν αυτή την πτυχή. Thank you. And now, Madam the Ευχαριστούμε κυρία Παντζέρη. Ευχαριστώ. Θα σταματήσω από εκεί που θα ξεκινήσω από εκεί από εκεί που σταματήσατε, για τα εξατομικευμένα δικαιώματα σε άδεια. Υπάρχει ε, το σημαντικό στοιχείο της ευελιξίας, δηλαδή αν κάποιος δεν πάρει για μιας ολόκληρη την άδεια, η οδηγία αποτείνει για τη γονική άδεια να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τα 12 έτη του παιδιού. Τέσσερα, τέσσερις μήνες, στη διάρκεια ζωής του παιδιού που μπορεί κανείς να παίρνει κατά τμήματα ε, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός αλλά και για τη δεύτερη παρατήρησή σα, σημαντικέ είναι οι αμοιβέ, ο μισθό. Δηλαδή, ε, το ίδιο και η άδεια φροντιστού. Είναι σημαντικό οι άδειε αυτέ να είναι αμοιβόμενε και να είναι σωστά αμοιβόμενε. Διότι η αμυστή άδεια δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Οι οικογένειε με χαμηλό εισόδιο δεν, μπορούν να, δεν θα μπορούν να τι πάρουν οι οικογένειε και θα αυξηθεί το χάσμα των μισθών ανδρών γυναικών. Πρέπει κάτι να κάνουν για να αντισταθμίσουν το εισόδημα ε, που θα λείπει από την οικογένεια και συνήθω είναι οι γυναίκε που τον πληρώνουν πάντα και μένουν εκτό δουλειά. Οπότε οι άδειε που είναι αμοιβόμενε είναι σημαντικέ. Είναι κάτι αυτό που προτείνει η Επιτροπή Ουσιμή Εφετηρία. Η πενθήμερη ε, άδεια είναι ήδη μια αρχή. Καλό θα ήταν να μπορεί κανεί να φτάσει ω τι 12. Αν κάποιο έχει μια χρόνια πάθηση, πηγαίνει συχνά για ιατρικά ραντεβού, θα μπορούσε να είναι μια μέρα το μήνα. Αλλά νομίζω ε, αυτή τη στιγμή είναι το μέγιστο στο οποίο θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Τώρα συμφωνώ και με του δυο σα όταν λέτε ότι η ανάγκη χαρτογράφηση είναι σημαντική. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη επακριβώ. Να δούμε τι υπάρχει για να σκεφτούμε στο μέλλον μακροπρόθεσμα τι ανάγκες υπάρχουν. Όμως θα πρέπει να είναι κάτι που θα το καταγράψουμε και οι γυναίκες δεν θα συμβάλλουν απλώς, μάλλον οι γυναίκες και οι άνδρες δεν θα συμβάλλουν απλώς στην κοινωνική ασφάλιση, γιατί βλέπετε, μου έρχεται αυτόματον από γυναίκες. Αυτές αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο των αδειών και της φροντίδας. Αλλά τέλος πάντων οι κοινωνικές ε, εισφορές να είναι και επιλογή. Να μην είναι τελευταίο καταφύγιο γιατί δεν υπάρχουν ε, άλλες λύσεις στην κοινότητα και στην κοινωνία. Οι γονεί και οι φροντιστέ εξαναγκάζονται να μείνουν εκτό αγορά εργασία τόσο καιρό που καταλήγουν όχι απλώ να μην μπορούν να έχουν μια κατάλληλη σύνταξη, αλλά δεν μπορούν να ξαναμπούν στην αγορά εργασία αν χρειαστεί να το θελήσουν. Οπότε, με το όριο, το προσδόκιμο ζωή διαρκώ να αυξάνεται, να ζουν όλο και περισσότερο οι άνθρωποι, είναι πιο δύσκολο να ξαναμπούν στην αγορά εργασία σε όποια ηλικία χρειαστεί. Τώρα, τελευταίο σχόλιο για τι υπηρεσίε. Και νομίζω ότι σημαντικό είναι παράλληλα με αυτά να σκεφτόμαστε και τα σχετική συζήτηση για τα διευθυντικά ταμεία μετά το 2020. Πρέπει να έχουμε μια εξάντερα σημότητα, 9,2, ε, για τις ε, κοινοτικές υπηρεσίες όπως έχουν ονομάσει, την ε, ίδρυμα, θεσμικοποίηση όπως έχει ονομαστεί σε όλου του κανονισμού για ταμεία πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η ισορροπία επαγγελματικού και γενικού βίου, οι υπηρεσίε φροντίδα και όλε οι σχετικέ υπηρεσίε παραμένουν μια καθοριστική προτεραιότητα. Διότι αν δεν παρέχουμε στι οικογένειε εργαλεία για να μπορούν να κάνουν τη σωστή επιλογή, οι οικογένειε δεν θα επιλέξουν τι θα κάνουν. Δεν θα μπορούν να επιλέξουν να κάνουν αυτό που θέλουν. Και ε, τελικά θα βρεθούν χωρί φροντιστέ. Πρέπει να είναι επιλογή των φροντιστών να είναι φροντιστέ. Και επιλογή του ανθρώπου που χρειάζεται βοήθεια φροντιστού να επιλέξει το φροντιστή του. Ιδίω ό,τι αφορά την τρίτη ηλικία και του γονεί. Έχω τόσα πολλά άλλα να πω, αλλά νομίζω θα σταματήσω εδώ για την ώρα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ όλου και όλε. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση και ένα πολύ σαφές μήνυμα. Ήταν συναρπαστικό το θέμα. Αποκαλύπτοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα στη φορολογία. Ήταν πραγματικά χρήσιμο. Και θα έλεγα και συγκινητική συζήτηση για μας αυτή την Επιτροπή. Για μας που είμαστε υπεύθυνοι για τα θέματα αυτά και για αυτές τις προτεραιότητες σας. Ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας και για τις παρατηρήσεις σας. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 12 Ιουλίου.